Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi ritengo opportuno iniziare, dare inizio ai lavori. Καλησπέρα. Ε, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους, ε, τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα τους ε, τρεις υποψήφιους. Πρώτο, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι έγκριση του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Να αναφερθώ στην ε, σημερινή διαδικασία. Η σημερινή συνεδρίαση είναι ανοιχτή σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τον ε, κανονά υπαριθμών 204. Ε, η, ε, η Επιτροπή Αναφορών έχει έξι υποψήφιους για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Μόνο τρεις υποψηφιώτε όμως γίνονται παραδεκτές σύμφωνα με τους κανόνες, με τι προποθέσει που αναφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε και σήμερα θα ακούσουμε τους ε, τρεις υποψήφιους με αλφαβητική σειρά, δηλαδή πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Βιτόριο Μπότολη, κατόπιν τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο και τέλος ε, τον κύριο Πιέρ Ιβ Μονέτ. Κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του μία ώρα. Μπορεί να παρουσιάσει καταρχήν την υποψηφιότητά του και κατόπιν να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών. Στο πρώτο τέταρτο θα ακούσουμε την παρουσίαση των υποψηφίων και μετά θα έχουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Και στο τέλος θα έχουμε και, μία, ε, ε, και ένα τέταρτο για τη διαδικασία Catch the Eye. Στην ιστοσελίδα μας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σε σχέση με, τις, με τη διαδικασία, οι, οι υποψήφοι που έγιναν δεκτοί και εκείνοι που δεν έγιναν δεκτοί. Επίσης έχουν εγγραφεί οι γραπτές ερωτήσεις και οι απαντήσεις των ιδίων. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με αυτή την ακρόαση. αλλά ήδη διαθέτουμε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε από αυτή την προκαταρκτική διαδικασία από τους μεμονωμένους υποψηφίους. Στο τέλος της σημερινής ακρόασης, των σημερινών ακροάσεων μάλλον, η Επιτροπή θα γνωμοδοτήσει και θα στείλει τη γνωμοδότηση στον πρόεδρο ε, του Κοινοβουλίου για να δούμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας και η τελική εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ε, άρχεται λοιπόν η ακρόαση και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπότολη να λάβει το λόγο. Non c'è. <laughs> Sì, sì. Sarà per arrivare. Θα, θα φτάνει τώρα, θα φτάνει τώρα. Μόλις φτάνει. Benvenuto. Ναι. Allora, gli diamo qualche minuto per... Ας του δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να καθίσει και επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μπότολη θα πρέπει να αρχίσει με μία παρουσίαση 15 λεπτών για να μας μιλήσει για τη δική του υποψηφιότητα και μετά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής. Honorable of Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία μετά τον πρώτο γύρο επιλογής να εμφανιστώ εδώ. Η εισαγωγή μου θα είναι σκόπιμα σύντομη. Από την πείρα μου έμαθα ότι η συζήτηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αναπτύξω τα θέματα που θα επιλέξετε εσείς για να αξιολογήσετε καλύτερα το πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά σας. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφήσουμε χώρο για οποιοδήποτε άλλο θέμα πιστεύετε ότι αξίζει την προσοχή σας. Αυτό είναι το μάθημα που έμαθα και που διδάσκω στους φοιτητές μου συνήθως ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς ως βουλευτές του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αυτής γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι προσβάσιμη η δημόσια διοίκηση και η πείρα μου στο θέμα αυτό φαίνεται από το βιογραφικό μου σημείωμα. Και το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας σημαίνει ότι θεωρήσατε παραδεκτή την υποψηφιότητά μου. Για οποιασδήποτε άλλες διευκρινήσεις βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Επιπλέον, Ήδη έχω απαντήσει γραπτός κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για σχετικά ζητήματα. Οι απαντήσεις μου αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες μου όσον αφορά τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή. Και για να έχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα. Υπάρχει όμως μια βασική αρχή μια θεμελιώδης αρχή την οποία θα πρέπει να επαναλάβω. Η επίσημη αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνεται στα συντάγματα όλων των κρατών μελών δεν αρκεί για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Η προστασία των δικαιωμάτων αυτών και μιλάω για την προστασία που παρέχει ο διαμεσολαβητή. Η προστασία αυτή δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλες τις περιφέρειες. Και υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ε, που έγινε στη Φλωρεντία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του φορέα αυτού, ε, είδαμε το εξής αποτέλεσμα, ότι σε πολλά κράτη-μέλη και σε πολλές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταργηθεί δια νόμου ο διαμεσολαβητής ή ο συνήγορος του πολίτη. Άλλοι δεν επαναδιορίστηκαν και άλλοι συνήγοροι του πολίτη έχουν αποκτήσει μικρότερη αξία, έχουν υποβαθμιστεί. Αυτά είναι γνωστά εδώ και καιρό και υπό το φως αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, ποιες είναι οι αιτίες της αρνητικής αυτής τάσης. Δεύτερον, τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, οι λόγοι είναι σαφείς σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει καθημερινές επαφές με τη δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το Κοινοβούλιο και η τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι δομές που έχουν καθιερωθεί για να υπάρχει διοίκηση μιας χώρας και για να υπάρχει ευημερία σε μια χώρα αυτή. Κάποια στιγμή όμως οι φορείς αυτοί ε, μπορεί να γίνουν σκοπός, να αποκτήσουν δική τους κυριαρχία και μάλιστα όχι μέσα στο συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο τους, αλλά με αξιώσεις για οικουμενικότητα. Τα... Οι φορείς αυτοί λοιπόν δεν προστατεύουν πάντα τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι γίνονται μέσω για τις ε, αρχές και έτσι οι αρχές αυτές δεν πληρούν πια τον ρόλο τους να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι σαφές ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις, διότι έχουν κοινή την ίδια υπηκότητα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίε που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία τους και για όλους τους συνηγόρους του πολίτη που συνδέονται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου να έχουν ένα σαφέ ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Σε περιπτώσεις λοιπόν σαφών διακρίσεων θα πετύχουμε με καλύτερη αποτελεσματικότητα εάν κατόπιν συμφωνίας με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή σας βρεθεί μια λύση. Γνωρίζω ότι μετά από 10 χρόνια αφοσίωσης στους πολίτες της χώρας μου και της περιφέρειάς μου. Η δέσμευση να παράσχω καλές υπηρεσίες είναι ακόμα πιο δυνατή. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Honorable President. Κυρία Πρόεδρε, ολοκλήρωσα την εισαγωγή μου. Νομίζω όμως ότι πολλές άλλες σημαντικές πτυχές μπορούν να αναλυθούν με περισσότερες λεπτομέρειες και θα προκύψουν από τις ερωτήσεις σας. Κυρία Πρόεδρε, Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα από εδώ και μπρος. Εξαιτίας της ευαίσθητης, ε, της φύσης αυτής της ακρόασης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, παρερμηνίες. Για να είμαι σίγουρος λοιπόν ότι εκφράζομαι σωστά, θα εκφραστώ στη μητρική μου γλώσσα στη συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Βιτόριο Μπότολη για την εισήγηση αυτή. Βεβαίως ε, θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον συγχαρούμε. Έχουν οι συνάδελφοι το λόγο και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σας έχουμε δώσει, ο καθένας μπορεί να παρέμβει δύο λεπτά. Η κυρία Γκρουνή είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Πότολη. Οι ερωτήσει μου. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του επόμενου διαμεσολαβητή, για την επόμενη δηλαδή θητεία, ποιες οι βελτιώσεις του ρόλου αυτού και κατά πόσο θα αλλάξει το οργανόγραμμα. Τι προβλέπουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να βελτιώσουν αυτή την υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των πολιτών και το ρόλο του Ombudsman όπως ορίζεται στις συνθήκες. Ποια είναι τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο θεσμών και θεσμικών οργάνων. Πώς ε, προβλέπετε την συνεργασία σας με την Επιτροπή Αναφορών, καθώς και με, τους, με τα άλλα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γκρουνή. Ο κύριος Ποσινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με καθηγητά. Να σας ρωτήσω το εξής. Τι προτείνετε για να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού, μάλλον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των εθνικών ομολόγων του σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ

πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των ε, εθνοτικών μειονοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα δικαιώματα φαίνεται να έχουν περιθωριοποιηθεί και ίσως η αιτία είναι ότι δεν θέλουμε να πλεχτούμε σε διάφορες συγκρούσεις που προκύπτουν από τα προβλήματα αυτά. Πολλοί ωστόσο πιστεύουν ότι τέτοιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να επιληθούν μέσω του διαλόγου δεν είναι καλή ιδέα να υποκρινόμαστε ότι αυτά τα προβλήματα, αυτές οι συγκρούσεις δεν υφίστανται. Ίσως λοιπόν ο διαμεσολαβητής θα μπορούσε να βοηθήσει, να συνδράμει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Και θα τη θέσω την ερώτηση αυτή και στους άλλους δύο υποψηφίους τα δικαιώματα των μειονοτήτων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο μέλλον θα τύχουν τις ίδιες αντιμετώπισης και ότι θα αντιμετωπιστούν ως συγκεκριμένο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, περιπτώσεις παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και άλλων τέτοιων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουγγαρία μεταξύ αυτών Πολλοί άνθρωποι λοιπόν στις χώρες αυτές έχουν την αίσθηση ότι τα δικαιώματα αυτά καταπατούνται και μάλιστα αγανακτούν γιατί δεν έχουν την αίσθηση ότι δίνεται προσοχή σε αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων. Ρωτάω λοιπόν το εξή. Συχνά οι εθνικές πολιτικές στρέφονται κατά των δικών μας πολιτικών, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κοινέ δεδελωμένες αξίες, οι οποίες εκφράζονται μέσω πολιτικών συγκεκριμένων. Τι γίνεται, έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για την ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, προκειμένου να μην έχουν οι πολίτες την αίσθηση ότι όντως υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την παραβίαση του δικαιώματος έκφρασης στην Ιταλία και τελικά αν θα αποφασιστεί ότι υπήρξε τέτοια παραβίαση, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες παραβιάσεις που αφορούν τεράστιες ομάδες του πληθυσμού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω ποια είναι η στάση σας έναντι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η στάση σας, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών σε ό,τι αφορά τις εθνικά δικαιώματα των μειονοτήτων. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση κύριε Μπότολη. Ε, ποιο ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσατε ως εθνικός διαμεσολαβητής και ε, με ποιον τρόπο προσπαθήσατε να το λύσετε και αν εκτιμάτε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ευρώπη ή τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζετε είναι εντελώς διαφορετικά ως Ευρωπαίος διαμεσολαβητής. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπότολη στην ε, σημερινή μας συνεδρία. Συζητώ συγγνώμη που δεν άκουσα όλη την παρουσίασή σας, άκουσα όμως το μεγαλύτερο μέρος. Τέσσερις ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Καταρχήν κύριε Μπότολη, ο κανονισμός περί διαφάνειας 1049 αναφέρεται στις διοικητικέ δραστηριότητες των θεσμικών οργάτων καθώ και στα κράτη-μέλη, καθώ και στο, στην εφαρμογή του ε, κοινοτικού νόμου. Υπάρχουν ε, κανόνες σε ευρωπαϊκό και επίπεδο και σε κρατικό επίπεδο που διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε τα δικαιώματα που ε, θεσπίζονται εκεί να προστατευτούν, ε, να μπορούν να εφαρμοστούν δηλαδή από τους πολίτες. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι πολύ πιο σύντομη. Εσείς προσωπικά πώς θα συμβάλλετε στη βελτίωση της ε, νοοτροπίας της υπηρεσίας, ε, των, του, της υπηρεσίας σας. Και τέλος, όσον αφορά αυτό που είπατε για το ότι οι υπηρεσίες γίνονται αυτοσκοπός ε, αντί να εξυπηρετούν το πολίτη, εσείς πώς θα διασφαλίσετε ο φορέας του διαμεσολαβητή να μην ε, καταλήξει έτσι και τέλος. Επειδή ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, συνήθως έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι θεσμός φιλικός προς, τον πολίτη, ιδιαίτερα υπό το φως ότι οι πολίτες συχνά δεν ξέρουν ε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ένα θεσμικό όργανο και στο άλλο. Πολλοί από εμά ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν συνειδητοποιούμε ότι ο πολίτης δεν γνωρίζει πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε. Θα επικεντρωθώ σε μία ερώτηση που βρίσκω ότι είναι ζωτική σημασία για τον διαμεσολαβητή. Το θέμα της καλής διακυβέρνησης και των καλών πρακτικών. τις οποίες θα πρέπει να εξετάζει ο διαμεσολαβητής πολίτης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχετε τη νομική βάση δύο νέα άρθρα σύμφωνα με τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την καλή διακυβέρνηση σε όλα τα θεσμικά όργανα. Εσείς πώς θα εφαρμόσετε αυτά τα άρθρα για να ισχύουν οι κανόνες αυτοί για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Μποτολή που τιμάτε με την παρουσία σας στη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Έχω την εντύπωση και την εντύπωση αυτή την έχουν και πολλοί ότι αλλάζουν πολλά πράγματα και με μεγάλες ταχύτητες στην εποχή μας και ιδιαίτερα στην Ευρώπη λόγω της μετανάστευσης, της ε, εμφυλοχωρήσεως ατόμων με διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικές, διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της ζωής. Ήδη πρόσφατα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί θέματος που αφορά την Ιταλική κυβέρνηση και την Ιταλική πολιτεία έκρινε το θέμα του Σταυρού ότι είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει στην ε, απομάκρυνση του Σταυρού από τα σχολεία, πράγμα το οποίο από τη μία πλευρά θίγει την πεποίθηση των αυτοχθόνων Ιταλών, οι οποίοι όπως ξέρουμε είναι καθολικοί χριστιανοί, και από την άλλη η διατήρησή του θίγει τους μετανάστες αριστρισκίας. Αυτό και μόνο το παράδειγμα δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διασφάλιση στην ισορροπία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς το ρόλο του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στη διασφάλιση της ισορροπίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια είναι τα όρια κατά την αποψή σας στη σύγκρουση των αγαθών και των αξιών τα οποία προανέφερα και τα οποία κατ' επέκταση είναι και πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Abbiamo finito Νομίζω ότι τελειώσαμε με τις ε, προγραμματισμένες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Βιτόριο Μπότολη για να απαντήσει και στη συνέχεια μετά τον πρώτο γύρο θα έχετε χρόνο μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye. Ο κύριος Μπότολη έχει το λόγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσω να απαντήσω πλήρως όσο το δυνατόν πληρέστερα σε αυτές τις ερωτήσεις σε σχέση με τον ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ιδιαίτερα πέρα από το θεσμό του Ομπούτσμαν γενικότερα. Βελτιώσεις. Ποιες βελτιώσεις θα ήθελε να εισαγάγει ο υποφαινόμενος εάν εκλεγεί ε, αύριο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Έχω ήδη δώσει απάντηση γραπτό στις γραπτές ερωτήσεις που μου έχει υποβάλει η Επιτροπή σας. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω αυτή την έννοια. Πιστεύουμε ότι σημαντικό δεν είναι μόνο να τονίσουμε το εύρος της δραστηριότητας και τα θεμέλια δημιουργίας αυτού του θεσμού σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιφέρειες, δηλαδή η αρρωγή προς τον πολίτη ως προς τις σχέσεις του με τη δημόσια διοίκηση. Όταν ο πολίτης θεωρεί ότι κάποιο δικαίωμά του έχει παραβιαστεί από τη δημόσια διοίκηση. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν αμφισημίες εδώ. Αυτό είναι και ο βασικός ρόλος του κάθε ombudsman σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια. Αλλά για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή νομίζω ότι υπάρχει μία άλλη εξίσου σημαντική πτυχή που μέχρι σήμερα δεν έχει τονιστεί επαρκώς. Αναφέρομαι στο άρθρο 5 του οργανογράμματος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπου αναφέρεται ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργαστεί με τους συναδέλφους και με τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνεργασία αυτή για μένα θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο ενεργός ρόλος του διαμεσολαβητή σε σχέση με τους άλλους ομπούτσμεν και τους θεσμούς που ασχολούνται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπα στην ε, εισήγησή μου, υπάρχουν περιφέρειες που βρίσκονται σε χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός διανόμου. Και για δεκάδες χρόνια οι διαμεσολαβητές δεν έχουν ε, ανανεωθεί, ας το πούμε έτσι. Δεν έχουν επανεκλεγεί. Και πολύ συχνά. Δεν μπορεί να γίνει πραγματική διαμεσολάβηση, δηλαδή ο Ombudsman περιορίζεται σε μία ταπέλα που υπάρχει σε ένα γραφείο. Άρα, τι εννοώ όταν λέω ότι ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει πολύ περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Τη στιγμή που ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο όλων των ombudsmen σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν λέω καθημερινά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία ανταλλαγή πληροφοριών και επαφές. Όλοι γνωρίζουν αυτή την κατάσταση της αποδυνάμωσης του θεσμού του Ombudsman σε επίπεδο ορισμένων κρατών ή κράτους γενικότερα. Εκεί λοιπόν που ο Ombudsman βλέπει ότι υπάρχει πρόδειλη παραβίαση δικαιωμάτων του πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει μία όχι μόνο ε, δικαιοδοτική εποπτεία, αλλά και μη δικαιοδοτική, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ κρατών και μεταξύ περιφερειών, κάτι το οποίο επισυμβαίνει σήμερα. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής που έρχεται σε επαφή με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με την Επιτροπή Αναφορών να καταγγέλει αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει δια την πανοκρουσίας. Θα πρέπει όμως αυτοδικαίως ο Ομπούτσμαν να μπορέσει να αντιδράσει και μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών. Τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι επικρίσεις, από όπου και αν προέρχονται, έτσι ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία λύτευση, ας πούμε. Ως προς τα δικαίωμα των μειονοτήτων. Μία από τις βασικές δραστηριότητες του Ombudsman στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών δεν αφορά γενικά την ε, προστασία υπό την αφαιρετική έννοια, αλλά τα δικαιώματα δεύτερης γενεάς, όπως έλεγε ο φιλόσοφος Μπόμπιο, δηλαδή τα ε, δικαιώματα της γυναίκας, των παιδιών, των ηλικιωμένων των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα των μειονοτήτων, διότι αυτές είναι οι πλέον ευάλωτες κατηγορίες που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, διότι η προστασία του πολίτη θα πρέπει να ευαισθητοποιείται προς αυτές τις ε, κατηγορίες, δηλαδή προς τους πιο αδύναμους και ευάλωτους της κοινωνίας μας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, γνωρίζετε ότι ορισμένα κράτη έχουν ε, θεσμοθετήσει τον Ombudsman, ο οποίος έχει αυτή την εξειδίκευση, δηλαδή την ε, υποστήριξη των μειονοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε Ombudsman θα πρέπει να προστατεύει τους πλέον ευάλωτους, τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες. ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Ομπούτσμαν, Δηλαδή στα 10 χρόνια δραστηριότητάς μου στην Επιτροπή του Βένετο σε σχέση με αρμοδιότητες που αφορούν ολόκληρη τη χώρα, δηλαδή την Ιταλία, διότι θα γνωρίζετε ότι στην Ιταλία ε, δεν υπάρχει ο θεσμός του εθνικού ομπούτσμαν. Εδώ και 50 χρόνια περιμένουμε ένα τέτοιο διορισμό. Υπάρχει λοιπόν περιφερειακός ομπούτσμαν, ο οποίος έχει αρμοδιότητες και στα πλαίσια του κεντρικού κράτους. Ποιο είναι το πιο μείζον πρόβλημα που αντιμετώπισε αυτή τη δεκαετία. Η απομόνωση. Η απομόνωση της περιφέρειας του Βένετο γιατί εμείς θέλαμε να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Από τις ε, αιτήσει το 2001 περάσαμε στις 11.000 πέρσι, που πιστοποιούνται από μία εποπτική αρχή. Και αυτό επειδή πέρα από τη βασική δραστηριότητα του Ombudsman προώθησα και μία επικοινωνιακή δραστηριότητα, διότι κανένα στην περιφέρεια, μιλώ για τους πολίτες της περιφέρειας, κανείς δεν γνώρισε ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Υπάρχει αυτό το πρόσωπο που ασχολείται με τους πολίτες. Άρα ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει ε, το πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό θα πρέπει να γίνει και από τους ακαδημαϊκούς κύκλους μέσω συναντήσεων, μέσω επαφών που υπάρχουν με όλες, όλους τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα που άπτονται του προβλήματος, αλλά επίσης θα πρέπει να ασχολείται και η περιφέρεια εκεί όπου υπάρχει αυτός ο θεσμός ο οποίος μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών τη στιγμή που υπάρχει παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων από την ε, δημόσια διοίκηση. Μίλησα για απομόνωση και απομονωτισμό. Στην περιφέρεια του Βένετο δεν υπάρχει μία επιτροπή, επιτροπή αναφορών. Άρα υπάρχει ένας μονοκρατισμός. Δηλαδή, θέλουμε βεβαίως να δώσουμε να υπάρχει μια ορατότητα, ένας ορίζοντας, έτσι ώστε να προωθούνται συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία για κάθε ombudsman είναι να έχει σημεία αναφοράς. Όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ε, τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το εφαλτήριο της Επιτροπής Αναφορών. Γι' αυτό προσπάθησα χρόνο με το χρόνο να δημιουργήσω μία τέτοια επιτροπή η οποία πλαισιώνεται από δημοτικούς συμβούλους ή περιφερειακούς συμβούλους που είχαν ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το θέμα της εποπτείας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών οι οποίοι με βοηθούσαν όχι μόνο να μην ε, θεωρήσω αυτόν απομονωμένο, αλλά με υποστήριξαν και σε όλες τις πρωτοβουλίες που έκρινα αναγκαίες για την ε, προστασία του πολίτη. Μου υποβλήθηκε και μία άλλη ερώτηση σε σχέση με την προσπελασιμότητα στην πληροφόρηση και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν. Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι ο βασικός νόμος, ο θεμελιώδης νόμος κάθε κράτους και κάθε περιφέρειας για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας. Γι' αυτό, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη μελέτησαν το θέμα και έθεσαν, έθεσαν επιτάπητος το θέμα της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και αρχεία. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένος από τον νόμο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως γνωρίζετε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως ε, δεν γίνεται κατάχρηση και σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, αλλά έχει δικαίωμα πρόσβαση σε όλα τα δημόσια έγγραφα. Άρα όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, διότι μέσω του Ombudsman οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα αν και την επαύριο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Δεν μπορούν να κοινοποιηθούν ούτε καν στον άμεσα ενδιαφερόμενο. Μπορεί όμως να μεσολαβήσει για να προασπίσει τα συμφέροντα του πολίτη και μέσα στα πλαίσια εγγράφων εμπιστευτικού χαρακτήρα. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειώσουμε και να συρρυκνώσουμε αυτή την ιερά αρχή της προσπελασιμότητας στα έγγραφα της δημόσιας διοίκησης. Ως προς τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα. που αυτοβούλος δρούν. Αυτό είναι και το θεμελιώδες ε, ζήτημα της δραστηριότητας του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Όλα τα συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανθρωποκεντρικά. Άρα το φυσικό πρόσωπο, τα φυσικά πρόσωπα είναι η πραγματική κυρίαρχη Η δημόσια διοίκηση στην ουσία υποστηρίζει αυτή την κυριαρχία του πολίτη και την υπηρετεί. Αλλά εάν αυτό το όργανο που υπηρετεί τον πολίτη λησμονεί ότι αυτή είναι η βασική του δραστηριότητα και υποχρέωση, τότε αυτό βούλος θα πρέπει ο πολίτης να τον επαναφέρει στην τάξη. Δηλαδή, η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πολίτη. Αυτό ορίζεται από όλα τα συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει οι δημόσιες διοικήσεις να ξεχνάνε τον πρωταρχικό τους ρόλο και να χρησιμοποιούν τους πολίτες μόνο όταν θα πρέπει οι πολίτες να εκλέξουν τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι ύψης της σημασίας για μας. Και δυστυχώς τα παραδείγματα που σας, έδειξα, που σας έδωσα πριν καταδεικνύουν ότι ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίστανται αυτά τα προβλήματα, διότι όταν σε μια Ιταλική περιφέρεια 20 χρόνια μετά από την δημιουργία του περιφερειακού ομπούτσμαν, όταν ένας νόμος κατάργησε αυτόν τον ομπούτσμαν μέσα σε 20 λεπτά και άρα γίνονται διακρίσεις εις βάρος αυτής της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιφέρειες της ίδιας της χώρας, αναρωτιέμαι κατά πόσο οι πολιτικοί που ψήφισαν αυτό το νόμο δεν ξέχασαν ότι αφαίρεσαν από τον πληθυσμό αυτό την δυνατότητα προστασίας των συμφερόντων του. Διότι αυτό είναι το βασικότερο σημείο. Δηλαδή, όχι μόνο να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα, αλλά να τα προστατεύσουμε και η προστασία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοτικής δραστηριότητας ή της εξοδικαστικής δραστηριότητας του Ombudsman. Αλλά σήμερα, σε αυτή τη στιγμή που ζούμε μια μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ποιοι είναι οι πολίτες οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν όταν παραβιάζεται ένα δικαίωμά τους, πώς μπορούν να υποστηρίξουν μία δράση και να προβούν σε μία προσφυγή. Τη στιγμή πρόκειται για μία δαπανηρή διαδικασία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ε, περιφέρεια του Βένετο, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε για μία βραδιπορία. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ombudsman μπορεί να δράσει με σπουδή και ανεξάρτητα, διότι δεν δεσμεύεται από ε, διοικητικές, διοικητικής μορφής περιορισμού, περιορισμούς. Υπάρχει μια φιλική σχέση, δηλαδή, έτσι ώστε να επιληθούν φιλικά και τα προβλήματα του πολίτη, εξοδικαστικά. Και εάν δεν επιληθούν, τότε ο Ομπούτσμαν οφείλει να παρεμβεί. Όχι φιλικά, αλλά με σπουδή και με την αυστηρότητα που επιβάλλεται. Τέλος, νομίζω ότι μια άλλη σημαντική πτυχή που επαναλαμβάνω είναι η πτυχή της επικοινωνίας και ιδιαίτερα ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, όχι μόνο τα κοινοβούλια, όχι μόνο οι πολιτικοί, αλλά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν αυτό το θεσμό και στις σχέσεις τους με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ξέρουν ότι έχουν έναν Ευρωπαίο Ομπούτσμαν που θα τους υπερασπιστεί πάντα. Αυτός ο θεσμός δεν είναι γνωστός σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Τον γνωρίζουν βεβαίως οι μικρές κοινωνίες και κοινότητας στην Ευρώπη είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, διότι ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής είναι μακριά από τα κράτη-μέλη, από τις πόλεις. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής να γίνει γνωστός σε όλα τα επίπεδα. Έφερα εδώ μαζί μου και ελπίζω να μην θεωρείτε ότι σας ε, δωροδοκώ ή σας διαφύρω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Είναι η τελευταία εργασία του δικού μου γραφείου. Είναι ένα, ε, όπως βλέπετε, ένα στην ουσία βιβλίο υπό μορφή κόμιξ. Σε 15 λεπτά ένα παιδί της μέσης εκπαίδευσης είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Υπάρχει το δικαίωμα της οικογένειας, το, τα εργασιακά δικαιώματα, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το καθεξής. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον πρώτο ομπουτσμαν της ιστορίας. Η Ρώμη έγινε res publica, δηλαδή θέμα όλων, υπόθεση όλων, διότι ο λαός επανήλθε στη Ρώμη όταν απέκτησε τον δικό του ομπούτσμαν μέσα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει γνωστοποίηση του ρόλου του ομπούτσμαν. Με συγχωρείτε εάν ε, δεν απάντησα σε όλα τα ερωτήματα, αλλά όταν μιλάει κανείς ε, ελεύθερα, ίσως καμιά φορά ε, παραβλέπει ορισμένες πτυχές. Αν ναι, να μου τις υπενθυμίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Ο κύριος Γκόμες ζήτησε το λόγο όμως τώρα μέσα στα πλαίσια του Catch the Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπότολη. Εν μέρει απαντήσατε ήδη στο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Θα ήθελα όμως να το πάω και λίγο παραπέρα. Είναι πολύ εντυπωσιακή η μέθοδό σας να διαφημίζετε τις δραστηριότητε σας ε, και τις ε, δραστηριότητε στα μαθήματά σας. Το, στην περιφέρεια του Βενέτο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για το διαμεσολαβητή. Πώς θα επιλέξετε να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο σε ό,τι αφορά την θέση, τον θεσμό αυτό. Ευχαριστώ. Κέλνερ. Thank Um, Ευχαριστώ να θέσω μία ερώτηση γιατί εξηγήσατε πώς βλέπετε το ρόλο σας έναντι των εθνικών συνηγόρων και διαμεσολαβητών και των πολιτών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η σχέση σας με τις άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως Europol, με την Τράπεζα Επενδύσεων Όλοι αυτοί οι θεσμοί σχετίζονται με τον πολίτη, αναφέρονται στον πολίτη. Πώ θέλετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ο ρόλο του διαμεσολαβητή σε σχέση με τι υπηρεσίε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπότολη, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη που έχασα την εισαγωγική σας ε, παρέμβαση. Ε, μια συμπληρωματική ερώτηση όμως που ταιριάζει πολύ με αυτή που μόλις ακούσαμε. Έχουμε την Επιτροπή Αναφορών, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, είναι και οι δύο φορείς που αποτελούν ένα σεισμογράφο για την Ευρώπη. Όταν πάει καλά η Ευρώπη δεν ε, λαμβάνουμε πολλές αναφορές, ενώ αντιστρόφως όταν δεν πάει καλά η Ευρώπη λαμβάνουμε πολλές. Εσείς είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει κατανοητή και αποδεχτού από τους πολίτες. Εμένα με ενδιαφέρει Πώς φαντάζεστε τη συνεργασία ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη συνεργασία αυτή και η δεύτερη ερώτηση, Πιο ωραίες είναι οι αναφορές όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τις, τους πολίτες. Μπορεί να μην μας ευχαριστούν οι πολίτες μετά, αλλά νιώθουμε την ε, προσωπική ικανοποίηση. Λαμβάνουμε όμως και αναφορές όπου νιώθουμε ότι θα, θα, θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παραθυράκια, κάποια κενά σε οδηγίες και κανονισμούς. Θα μπορούσατε να φανταστείτε μια κατάσταση όπου να επισημαίνετε στο Κοινοβούλιο ότι εδώ υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ε, Ίσως θέλετε ε, μια διευκρίνηση γιατί έχετε ήδη παρέμβει. Ε, επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά με τα όρια τα οποία ε, τάσσονται στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και επειδή πιστεύω ότι η αποτελεσματικότητα ενός θεσμού έχει σημασία και όχι η ρομαντική περιγραφή του θεσμού. Θα ήθελα να έχω την άποψη του κυρίου Βότολη πάνω στο θέμα του ποια είναι η άποψή του και πώς βλέπει το ρόλο του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στη διασφάλιση της ισορροπίας αυτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια τα όρια στη σύγκρουση καθηκόντων και στη σύγκρουση αγαθών και αξιών η οποία παρουσιάζεται στις μέρες μας όλο και πιο έντονη. Εάν δούμε τη ρομαντική άποψη του θέματος, φτιάχνουμε ένα θεσμό ο οποίος είναι απογυμνωμένος. Εγώ πιστεύω ότι ο Όμπουσμαν πρέπει να γίνει ουσιαστικός θεσμός, διότι η δικαιοσύνη αργεί. Ο Όμπουσμαν σαν εξοδικαστική λύση προβλημάτων, ιδιαίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει και ταχύτητα να έχει και αποτελεσματικότητα και ρεαλισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου προσδιορίσετε κατά την άποψή σας τα όρια των καθη... της συγκρούσεως καθηκόντων τα οποία ως ημέρα έρχονται στο φως της πραγματικότητας της ευρωπαϊκής. Λοιπόν, να σας ε, ρωτήσω το εξής για να αποφύγουμε τις παρανοήσεις γιατί είτε η Επιτροπή, μάλλον και η Επιτροπή μας και ο Διαμεσολαβητής, ε, δεν είμαστε ο Άγιος Βασίλης. Είναι σημαντικό να περιοριστούμε στις αρμοδιότητες μας. Να παραμείνουμε στο πεδίο αρμοδιότητων του διαμεσολαβητή. Μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα των μειονοτήτων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από όσο ξέρω όμως δεν έχει αρμοδιότητες ο διαμεσολαβητής σε αυτά τα πεδία. Σα παρακαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη ότι είναι καλά ορισμένε αυτέ οι αρμοδιότητε και θα πρέπει σε αυτέ να αναφερόμαστε, στις αρμοδιότητε δηλαδή του διαμεσολαβητή. Σωστό κύριε Μποσινάρου, διότι αυτές οι αξιολογήσεις ε, αφορούν πολιτικές πτυχές που δεν σχετίζονται με, με το λειτουργήμα του διαμεσολαβητή. Εγώ εξαιτία του ρόλου μου θα ήθελα να ζητήσω στον κύριο Μπότολη να απαντήσει, έχει το λόγο για ακόμα 7 λεπτά και να μας πει συγκεκριμένα πώς θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών. Ποιες, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ενδεχόμενοι μηχανισμοί, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι πιο παραγωγική και η Επιτροπή Αναφορών αλλά και ο θεσμός του Ombudsman για να προασπίσουν την προστασία, την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Έχει το λόγο κύριε Μπότολη. Νομίζω ότι μίλησα για τον, ως προς το επικοινωνιακό σκέλος. Τα θεσμικά όργανα πολλαπλασιάζονται. Υπάρχει αυτός ο πολλαπλασιαστικός παράγων και τα μέσα κοινοποίησης των αλλαγών στο, στο, στους πληθυσμούς ε, αποκλίνουν. Δηλαδή ένα διαφημιστικό σποτ υπομορφή καρτούν μπορεί να είναι πιο αποδοτικό υπομορφή κινούμενων σχεδίων καθώς και μία σειρά επεισοδίων όπου ο πολίτης μπορούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικός με τον ομπούτσμαν και να υποβάλει το ερώτημά του. Διαπιστώσαμε την επομένη ότι υπήρχαν όλο ένα και περισσότερες αιτήσει στη συνέχεια μέσω σχολείων να έρθουμε σε επαφή με τους ε, επιθεωρητές εκπαίδευσης, να προωθήσουμε δελτία, να έρθουμε σε επαφή με επαγγελματικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα μορφών, χρειάζεται και φαντασία. Θα πρέπει όμως να υπάρχει η βασική δέσμευση, ότι δηλαδή ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να περιορίζεται στη δραστηριότητά του, στη διοικητική του δραστηριότητα. Θα πρέπει να διαδίδει αυτές τις γνώσεις, γνώσεις που αφορούν και το γνωστικό του αντικείμενο. Τώρα, ως προς τη σχέση ε, με τους άλλους φορείς. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση Όσο περισσότερο συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, τόσο τα θεσμικά όργανα θα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Ombudsman διαδραματίζει ρόλο εισαγγελέα ή έχει ανακριτικό ρόλο. Τη στιγμή που η συνεργασία αυτή δείξει ότι υπάρχει πρόδειλη παραβίαση ενός δικαιώματος που δεν αναγνωρίζει η δημόσια διοίκηση, που παραβίασε το δικαίωμα του πολίτη, βεβαίως θα αλλάξει και η θέση του διαμεσολαβητή. Δεν θα είναι ο μελιστάλαχτος διαμεσολαβητής, αλλά θα παρέμβει δυναμικά για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη οι σχέσεις τώρα ως προς σχέση με την Επιτροπή Αναφορών. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Όταν σας είπα γιατί αισθάνομαι, αισθανόμουν μόνος στη δική μου περιφέρεια, γιατί δεν πλαισιωνόμουν από μια Επιτροπή Αναφορών. Αυτό, αυτό που έχει σημασία είναι η αγαστή συνεργασία με ένα τέτοιο όργανο. έχει μεγάλη σημασία ο πολλαπλασιαστικός ρόλος που μπορεί να ε, εξευρεθεί και μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών. Γι' αυτό μιλάμε για μονοκρατισμό του Ombudsman, αλλά μέσα στα πλαίσια της ε, πλαισίου αυτής από την Επιτροπή Αναφορών υπάρχει ένας συλλογικός χαρακτήρας διοίκησης. Άρα μέγιστη δυνατή συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά ιδιαίτερα με την Επιτροπή Αναφορών. Επίσης, στην τελευταία παρέμβαση ε, ελέγχθη ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε πολιτική χρειά στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά να μιλήσουμε για τα προνόμια και τα καθήκοντα του ομπουτσμαν. Μα ένας ε, ομπουτσμαν δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την πεμπτουσία της, ε, του ρόλου του που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει μεγάλη σημασία όταν βλέπει ότι υπάρχουν διακρίσεις ή όταν γίνεται παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Εγώ, ε, εάν προστατεύω τον πολίτη και αν ο πολίτης έρθει σε μένα και μου πει ότι με ζημίωσε η δημόσια διοίκηση κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ ακούω τον πολίτη, προσπαθώ να επιλύσω το πρόβλημά του. Που είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Πώς να μην ασχοληθώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν όλους τους λαούς και όλες τις δημόσιες διοικήσεις. Ο συνήγορος του πολίτη είναι το κλαδί ενός μεγάλου δέντρου. Το δέντρο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κλαδί ενός γερού δέντρου και δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον κορμό και στις ρίζες. Διαφορετικά ο Ombudsman δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όταν λοιπόν λέω ότι διαμέσου αυτού του δικτύου θα δράσουμε, θα συνεργαστούμε και ο καθένας από μας γνωρίζει σε πραγματικά χρόνο τι συμβαίνει σε άλλα σημεία της Ευρώπης και μέσω της στενής συνεργασίας με την Επιτροπή Αναφορών έτσι ώστε να στυλιτεύσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πολιτική χρειά σε όλα αυτά. Ο συνήγορος του πολίτη ορίζει τις περιπτώσεις και τις περιστάσεις που πρέπει να στυλιτεύσουμε. Και στη γραπτή μου απάντηση αναφέρθηκα και στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αναφορών. Θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση, συνεχής διαβούλευση, δηλαδή αν η Επιτροπή Αναφορών δεν επιτρέπει δεν επιτρέπει την παρέμβαση του Ευρωπαίου ε, Διαμεσολαβητή, δεν μπορεί να παρέμβει. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί συνέβη πρόσφατα σε μια περιφέρεια της χώρας μας. Ο, με συγχωρείτε, θα πρέπει να κλείνετε ο πρόεδρος, μάλλον ο Ευρωπαίος Διομεσολαβητής παρενέβη στην, ε, σε επίπεδο περιφέρειας που προήγει αυτό το νόμο, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του νόμου, ο οποίος κατάργησε το συνήγορο του πολίτη σε αυτή την περιφέρεια της ε, Ιταλίας. Εν πάση περιπτώσει, ο οποιοδήποτε ομπούτσμαν θα πρέπει να προστατεύει κάθε περίπτωση τη στιγμή που παραβιάζονται τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε πολίτη. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Μπότολη. Σε αυτό το σημείο και ενώ θα αποχωρήσει ο κύριος Μπότολη, θα ήθελα ο κύριος Διαμαντούρος να λάβει θέση για να προχωρήσουμε με τη δεύτερη ακρόαση. Allora, Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, καλοσύνη σας και για την πρόσκλησή σας. Ε, θα συνεχίσω στα αγγλικά με την άδειά σας. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσω το όραμά μου και τις ε, φιλοδοξίες μου για τη θέση του ε, Ευρωπαίου Διάσημου Μεσολαβητή. Έχω υποβάλει σε 23 γλώσσες ε, το βιογραφικό μου σημείωμα, το οποίο τονίζει τα βασικά προσόντα που φέρνω στη θέση αυτή. Καταρχήν η επαγγελματική μου εμπειρία ως συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ως Ευρωπαίο Μεσολαβητή μετά τον Απρίλιο του 2003 Τέλος, ε, την ε, ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 225 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα 27 κράτη-μέλη που ε, επιβεβαίωσαν την υποψηφιότητά μου για να ξαναυποβάλω υποψηφιότητα. Αποτελεί τιμή για μένα το γεγονός ότι τόσοι βουλευτές από τόσες διαφορετικές πολιτικές ομάδες με υποστήριξαν μια τέτοια ευρεία υποστήριξη αποτελεί ε, μια σημαντική ε, υποστήριξη για τον ε, νομιμοποίηση για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη. Διαμεσολαβητή θα ήθελα του Ευρωπαίου πολίτη, συγγνώμη. Θα ήθελα να σας αναφέρω τα επιτεύγματά μου. Καταρχήν, μια πιο αποτελεσματική προσφυγή για τους πολίτες σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και η μεγαλύτερη διαφάνεια. Με τις ε, έρευνες πρωτοβουλία μας αλλά και με τις ε, απαντήσεις στις προσφυγές έχω βελτιώσει τις βέλτιστες πρακτικές με τις ετήσιες εκθέσεις μου όπου δίνω παραδείγματα της ε, καλής διακυβέρνησης Έχουμε λύσει ε, προβλήματα ε, καθυστερημένων πληρωμών, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ε, μεμονωμένους πολίτες. Επίσης, έχουμε ασχοληθεί με την υπερβολική γραφειοκρατία, ιδιαίτερα εις βάρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε βελτιώσει την διαδικασία επιλογής της ΕΠΣΟ, και ως αποτέλεσμα το 2008 40% λιγότερες προσφυγές κατά της έπσο είχαμε από ότι το 2007. Έπεισα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνονται σε αιτήματα των πολιτών και να λαμβάνουν υπόψη την προοπτική του πολίτη όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Επίσης έκανα αυτά που έλεγα. Ε, προσπάθησα να ε, θέσω ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά την υπηρεσία προς τον πολίτη, ιδιαίτερα η υιοθέτηση. Υιοθέτησα νέο σαφή μορφότυπο για τις αποφάσεις και ε, επίσης εκπαιδεύσαμε στα απλά αγγλικά το προσωπικό μας για να είναι πιο κατανοητές οι αποφάσεις. Πάνω από 200 ομιλίες έκανα για να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους ε, όσον αφορά τις προσφυγές. Επίσης, είχαμε καλή ε, διακυβέρνηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό στην οργάνωση του φορέα μας. Ε, αναδιοργανώσαμε την ιστοθέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για να είναι ελκυστική και κατανοητή σε 23 γλώσσες. Την ετήσια έκθεση την κάναμε πιο σύντομη, πιο επικεντρωμένη στα βασικά θέματα και πιο φιλική προς αναγνώστη. Επίσης, ε, βελτίωσα την ε, πρόσβαση στις πρόσφυγες για τους πολίτες ε, και σε επίπεδο ένωσης χρησιμοποίησαμε πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες. Έχουμε συντομεύσει το χρόνο για τη λύση των προσφυγών και έχουμε εκδώσει έναν οδηγό που βοηθάει τους ε, πολίτες, στις ε, επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο οδηγός αυτός ήδη έχει χρησιμοποιηθεί από πάνω από 24.000 πολίτες από ε, την έκδοσή του φέτος τον Ιανουάριο. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης. Η τράπεζα έχει βελτιώσει το σύστημα προσφυγών της Επίσης, ε, ξεκινήσαμε ετήσιες ε, μελέτες ε, και χρησιμοποίησα τις ενισχυμένες αρμοδιότητες που μου έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε επίπεδο κρατών μελών συνεργάστηκα με εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές για να ενισχύσω το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες στις διάφορες περιφέρειες. Η συνεργασία αυτή βελτιώθηκε με πάνω από 100 επισκέψεις σε όλα τα κράτη-μέλη, όπου συνάντησα πολίτες, δημόσιες διοικήσεις, την κοινωνία των πολιτών, μέλη των κυβερνήσεων και το δικαστικό σώμα. Πρόθεσα την υιοθέτηση μιας δήλωσης από όλα τα μέλη του δικτύου όσον αφορά την, τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες. Βελτίωσα τις ε, υπηρεσίες συμβουλών προς τους εθνικούς συνηγόρους του πολίτη που έχουν απορίες σχετικά με το ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ερμηνεία τους. Έτσι βοηθάμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σωστά το ε, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ενθαρρύναμε την καλή επικοινωνία ανάμεσα στους διαφόρους συνηγόρους του πολίτη και το δίκτυο Solvit. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1041 του 2001, προωθήσαμε την ε, διαφάνεια, βελτιώσαμε την πρόσβαση των πολιτών στα ε, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν ε, συμφωνία και μάλλον υπογράψαμε μνημόνιο κατανόησης με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την προστασία των δεδομένων αναπτύξαμε επαφές με εθνικούς ε, επιτρόπους για την πληροφόρηση στα κράτη-μέλη, ε, ε, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία. Γενικά κατάφερα να βοηθήσω το 80% των ανθρώπων που προσέφηκαν σε μένα είτε άμεσα είτε παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να στραφούν σε περίπτωση που δεν μπορούσα να ξεκινήσω εγώ έρευνα οι δραστηριότητες πρωτοβουλίας μου ε, ε, ε, βοήθησαν στο διπλασιασμό της κάλυψης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή και στην υποβολή σημαντικών υποθέσεων για θέματα αρχής, θέματα που είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα υπεράσπισης, την κατάχρηση εξουσίας κλπ. Σύμφωνα με το Ευρωμάτρο του Μαΐου 2008, το 38% των Ευρωπαϊκών πολιτών γνωρίζουν τι είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Έχουν ακουστά το Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό νούμερο, δεδομένου ότι η εντολή του διαμεσολαβητή περιορίζεται στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υπηρεσίε του. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρί ε, την συνεργασία του ε, Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο μου έδωσε το δυναμικό που χρειαζόμουν για να κάνω τη δουλειά μου και η Επιτροπή σας ασχολήθηκε ε, αποτελεσματικά με θέματα στα οποία επέστρεψα την προσοχή σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ειδικέ εκθέσεις που θεώρησα ότι είναι απαραίτητο να υποβάλω. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σίγουρα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά θεωρούνται απόμακρα και απρόσωπα μία απρόσωπη γραφειοκρατία. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ε, συμφωνία μεταξύ μας ότι η διατήρηση υψηλής ποιότητας ε, στην ε, διοικητική πρακτική όχι μόνο θα ωφελήσει τους πολίτες, αλλά θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αυτά. Είμαι περήφανος για τα αποτέλεσματα που έχω πετύχει ως διαμεσολαβητής, ωστόσο γνωρίζω ότι Υπάρχουν πολλά που πρέπει και μπορούν να γίνουν ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν απόλυτα τα δικαιώματά τους ε, και πώς μπορούν να τα ασκήσουν. Είναι σαφές από τις απαντήσεις ε, των θεσμικών ε, οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης στις έρευνές μου ότι ήδη υπάρχει υψηλό επίπεδο διοικητικής πρακτικής. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων για την ε, κακή διαχείριση είναι πολύ λίγε. Μόνο 16 ειδικέ εκθέσεις έπρεπε να υποβάλει ο διαμεσολαβητής σε 14 χρόνια λειτουργία του. Ωστόσο, οι βελτιώσει μπορούν και πρέπει να γίνουν από τι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ε, δημιουργηθεί μια κουλτούρα υπηρεσίας προς τον πολίτη. Ένας τέτοιο στόχο μπορεί να βοηθηθεί από έναν διαμεσολαβητή που είναι απόλυτα ανεξάρτητο και δίκαιο και αμερόληπτος. Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο έχω επιδιώξει συστηματικά στα χρόνια που, της θητείας μου και που θα συνεχίσω να επιδιώκω εάν επανεκλεγώ. Όπως ε, ήδη ε, έχω πει στις ε, απαντήσεις μου σε ερωτήσεις που στείλατε σε όλους τους υποψηφίους και όπως ήδη έχει, αναγράφεται στην ιστοθέση του διαμεσολαβητή, ε, υπάρχουν τρεις προτεραιότητες ε, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει τον πολίτη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχυθεί η κουλτούρα υπηρεσία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της θέσης του ε, Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω τις ιδέες που ανέφερα στις γραπτές μου απαντήσεις. Κύριο στόχο των ε, θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι να καταστήσουν επιτυχία την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα και να ε, κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πολίτη. Η συμβολή του διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι ότι οι πολίτες θα αποφελούνται από την καλή διοίκηση και ότι θα γνωρίζουν τις διατάξεις της συνθήκη όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, να μπορούν να προσφύγουν στον διαμεσολαβητή μεσολαβητή ή στο κοινοβούλιο ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Στοχεύω να επικαιροποιήσω τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής ε, Διοικητικής ε, Πρακτικής ε, υπό το φως των βέλτιστων πρακτικών που έχει αναπτύξει ο διαμεσολαβητής και άλλοι και την ε, διοικητική νομολογία και την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ώστε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν τον κώδικα αυτό και να τον ακολουθούν όσο γίνεται. Θέλουμε να αναπτύξουμε την ε, δυνατότητα ερευνών πρωτοβουλίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα άτυπο δίκτυο καλής διοίκησης, να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές, να παρέχουμε κατάρτιση, να συνεργαζόμαστε στενά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους φορείς της, ώστε να διασφαλίσουμε τις φιλικές λύσεις. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή αυτή και με το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Επιπλέον, προτείνω στο νομοθετικό διάλογο να έχω μια πιο ε, ισχυρή θέση, να παρεμβαίνω στις δημόσιες συζητήσεις όσον αφορά την προτινόμενη νομοθεσία για θέματα που αφορούν τον ε, διαμεσολαβητή, όπως είναι ε, ο κανονισμός για τον Όλαφ, ο δημοσιονομικός κανονισμός κλπ. Εάν με επανεκλέξετε, προτείνω να κάνω τα εξής. Να ενισχύσω τις ε, επαφές με εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, και την, ε, και την καλύτερη πληροφόρηση. Να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για την οργάνωση εκδηλώσεων που θα χρησιμοποιούν την εμπειρία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επίσης, ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους φορείς πληροφόρηση του Κοινοβουλίου για να ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες. Τακτικά να οργανώνουμε εκδηλώσεις ε, μαζί με, σε συνεργασία με ενδιαφερομένους ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δημιουργήσουμε ένα, φόρουμ, ένα συνεχές φόρουμ για διάλογο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ιστοθέσεις ε, κοινωνικής δικτύωσης ε, για να ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τους πολίτες. Και τέλος θέλουμε να βελτιώσουμε την γνωστική βάση των του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών ε, και Παρομοίων Φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η βελτίωση της ποιότητας ε, της διοίκησης προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη πάντα ήταν βασικός μου στόχος. Εάν με επανεκλέξετε θα υιοθετήσω ένα στρατηγικό σχέδιο για τη θέση του διαμεσολαβητή που θα έχει ως light motif ε, την εξή δήλωση. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει τις δίκαιες λύσεις σε προσφυγές κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνει την διαφάνεια και προωθεί μια ε, διοικητική κουλτούρα της υπηρεσίας. Θέλει να βελτιώσει την ε, εμπιστοσύνη μέσα από τον διάλογο με τους, με πολίτες ε, και την... τον διάλογο μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, οδηγηθούμε σε καλύτερα πρότυπα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε μια διοίκηση με ανθρώπινο πρόσωπο που να είναι αφοσιωμένη στην ε, εξυπηρέτηση των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Τώρα ανοίγει η συζήτηση. Γκρουνή, πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Διαμαντούρο. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις που σας υπέβαλα γραπτός, γιατί μας τις ε, ανακεφαλώσατε και στην απάντησή σας, στην εισήγησή σας μάλλον τώρα. Μέσα στα πλαίσια της θητείας σας θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα θέλατε να εφαρμόσετε κάτι που δεν μπορέσατε μέχρι τούδε. Έχετε νέους στόχους πραγμάτωση. Δεν φοβόσαστε να έχετε μία θητεία που θα είναι μία θητεία η οποία θα είναι μία παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και πώς βλέπετε τη συνεργασία σας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ευρωπαίη Δημοσιολάβητη. είναι μεγάλη μου χαρά και ιδιαίτερο πλεονέκτημά μου να σας καλωσορίσω εδώ στην ακρόαση αυτή. Με στενή συνεργασία με την Επιτροπή μας του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, οι πολίτες μπορούν πλέον να δουν καλύτερα ποια είναι η διαφορά μεταξύ καλής και κακής διαχείρισης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε για ένα κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης των αναφορών προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διαμαντούρε, να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα επαναληφθώ ως ένα βαθμό αλλά στις γραπτές σας, στη γραπτή σας εισήγηση, αλλά και στα προφορικά σας σχόλια, περιλαμβάνεται ένα σημείο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν το βρήκα όμως την παρουσίασή σας στο σημείο αυτό, το θέμα των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων. Δεν ήμουν ίσως σαφής προηγουμένως, δεν έδωσα παραδείγματα, θα δώσω παραδείγματα. Μπορεί σε ένα κάποιο κράτος μέλος ο νόμος να προβλέπει ότι οι εθνικές ε, μειονότητες δεν μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουν την εθνική τους γλώσσα. Την γλώσσα τους. Μιλάμε για μια συλλογική παραβίαση δικαιωμάτων. Αλλά και παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου που προκαλεί προσωπικά πόνο σε κάθε άτομο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, τι μπορείτε να κάνετε εσείς, τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει γενικότερα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Πώς μπορούμε να βρούμε μια έναν ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών αυτών. Χωρίς να αγνοούμε τις παραβιάσεις αυτές, χωρίς να κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, πρόκειται για παραβιάσεις που επηρεάζουν τόσο ολόκληρες ομάδες, αλλά και μεμονωμένα άτομα του πληθυσμού. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και περισσότερο σε πιο αφρημένο επίπεδο, αν θέλετε. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί θέλουμε να επιλύσουμε συγκεκριμένες διαφορές, αλλά και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται μια αίσθηση αγανάκτησης, ότι κάποιους ανθρώπους τους παρατάμε δηλαδή. Και έχει ο κόσμος την αίσθηση ότι εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του πρόβλημα, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Αν και η παραβίαση των ατομικών αυτών δικαιωμάτων σημαίνει και η παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για την αξιοπρέπεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, σας ρωτώ, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις και πώς θα καταργήσουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά τα οποία εφαρμόζονται και σε πιο γενικό επίπεδο. Εσείς, πώς μπορείτε ως διαμεσολαβητής να εξασφαλίσετε ότι θα εφταμιγραμμιστούν οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες για να μην υπάρχουν κρίσεις δομής. Thank you very much. Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντούρε, κυρία Γκέντς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ συνοπτική και μιλήσατε και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Σας ευχαριστώ γιατί ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Ποιες αλλαγές δηλαδή οραματίζεστε μετά την συνθήκη της Λισαβόνας και την ε, εφαρμογή της. Απαντήσατε όμως το ερώτημα αυτό, δεν χρειάζεται να το ξαναθέσω. Μία άλλη ερώτηση όμως, την οποία έθεσα και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Μειώσατε σημαντικά τη διάρκεια χρόνου που αφιερώνεται στην απάντηση ερωτημάτων των πολιτών. Είναι ευαίσθητο θέμα αυτό, ξέρετε, γιατί αν ο κόσμος έχει κάποια ερώτηση, θέλει να απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το θέμα της διάρκειας απάντησης των ερωτήσεων αυτών, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ανακύπτει συχνά. Η κυρία... Wallace. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Διαμαντούρο για την πολύ θετική παρουσίασή σας σε δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν, όλοι αναγνωρίζουμε την αφοσίωσή σας ε, στην ε, κουλτούρα υπηρεσία στα θεσμικά όργανα. Πολλοί όμως ανησυχούμε ακόμα ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμετώπιοι με μια πληθώρα μερών όπου μπορούν να στραφούν, μπορούν ε, να στείλουν αναφορά στο κοινοβούλιο, μπορούν να στραφούν σε εσά, ε, μπορούν να ψάξουν στο Solvit, μπορούν να ε, έρθουν σε επαφή με την Κομισιόν. Όλα αυτά μπερδεύουν τους πολίτες. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για το, πού πρέπει να στραφούν. Ε, έχει αναφερθεί η λύση της ενιαίας στηρίδας ή μιας κοινή πύλης. Τι πιστεύετε εσείς. Δεύτερον, η μιας κοινης πυλης τι πιστευετε εσεις δευτερον η λισαβονα θα σημαίνει ότι το Συμβούλιο θα είναι ένα πολύ πιο σταθερό θεσμικό όργανο, θα παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ήταν όμως υπόδειγμα διαφάνεια τα τελευταία χρόνια. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό και τι θα γίνει με τα κοινοβούλια των κρατών μελών που πλέον θα συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Προβλέπετε η ειδική σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. και πώς βλέπετε τον πιθανό τους ρόλο ως νέο θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας και την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πολλές από τις ερωτήσεις μας μοιάζουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα έχουμε δύο νέα άρθρα που προσφέρουν νομική βάση για βελτίωση της διακυβέρνησης στα θεσμικά όργανα. Μιλήσατε γι' αυτό. Θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα τι θα κάνετε γι' αυτό. Θα έχουμε κανόνες που να επιβάλλουν την καλύτερη διακυβέρνηση και επίσης όσον αφορά την παρακολούθηση των διαφόρων φορέων και θεσμικών οργάνων. Πώς θα βελτιώσετε την παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Διότι νομίζω ότι αυτό θέλουμε να κάνετε και αυτό είναι πολύ κοντά στους πολίτες, διότι πολύ συχνά έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριο Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το βιογραφικό σας και την ε, πολύ ε, ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Φαίνεται ότι ε, θέλετε πολύ να συνεχίσετε τη δουλειά που έχετε κάνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι θεωρείτε την, ποια θεωρείτε την καλύτερη μεμονωμένη απόφασή σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας και δεύτερον ποια μεμονωμένη δράση ή απόφαση ε, έχετε μετανιώσει και θα ήθελα να ξέρω γιατί και στις δύο περιπτώσεις. Ε, στην γραπτή σας απάντηση αναφερόσαστε στην ε, θεσμοποίηση της παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται από τον διαμεσολαβητή σε υποθέσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι λάβαμε απάντηση σε αυτό. Αν απαντήσατε, έχασα, θα ήθελα να αναπτύξετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητώντα την έκθεση της κυρίας Παλιαδέλη που είναι στο Βήμα, είναι στο Προεδρείο, ε, να, εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε κατά τη γνώμη μου θετικά το έργο του κυρίου Διαμαντούρου. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του και για το έργο του και αξιοποιώντα τη σημερινή παρουσία του εδώ θα ήθελα να του υποβάλω ορισμένα ερωτήματα. Το πρώτο, από την εμπειρία του, τι προβλήματα συνάντησε με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές και πώς τα έλυσε. Πώς πρέπει να λύνονται τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο, μιλάει στη γραπτή απάντηση για την ανάγκη να προαχθεί και να παγιωθεί μια νοοτροπία εξυπηρέτηση του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Δίκηση. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη, ένας δύσκολος στόχος. Όταν μάλιστα αναφέρεσαι σε όργανα πολυσχηδή, αδιαφανή και κατά βάση μη ερετά. Εδώ κύριε Διαμαντούρο τι θα κάνουμε. Και το τρίτο για να μπορεί να προασπίσει, να, να γνωρίζει και να προασπίσει τα δικαιώματά του ο πολίτης, πρέπει να τα γνωρίζει. Αλλά κατά την εκτίμησή μου, η συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά και ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Επομένω, εδώ ποια κατά τη γνώμη σα, ποιε ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σα, για να μπορεί να γνωρίζει καταρχήν ο πολίτη τα δικαιώματά του, για να τα προασπίσει και να παραπέμπει ή να αναφέρεται σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαλαβράκο. Κύριε Διαμαντούρο, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω και εγώ τον απολογισμό του έργου σα και την έκθεση τη κυρία Παλιάδέλη, και πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Οφείλω να το ομολογήσω. Όμω από αύριο αρχίζει μια καινούρια εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόζεται η συνθήκη τη Λισαβόνα και τα ίδια προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν και για το κοινοβούλιο αυτό Τη αποτελεσματικότητα και τη ουσιαστική δηλαδή παρεμβάσεω του στα βήματα τη κοινότητα, παρουσιάζονται για όλου του παρεπόμενου θεσμού μεταξύ των οποίων είναι και ο θεσμό του Όμπουσμαν. Πρέπει να διατηρηθούν ορισμένε, πιστεύω αποτελεσματικέ ε, και να διασφαλιστούν ορισμένε αποτελεσματικέ παρεμβάσει που αφορούν τόσο εμά όσο και το θεσμό, του Όμπουσμαν. Έχετε επισημάνει εσεί πως ο θεσμός του Ευρωπαίου Μεσολαβητή εν ώψη της συνθήκης της Λισαβόνας και της εφαρμογής της θα γίνει πιο αποτελεσματικός για να μιλάμε πλέον σε ρεαλιστικό επίπεδο και όχι σε ένα επίπεδο ευχών ή ένα επίπεδο υπερβολικής ευγενίας και μη ρεαλισμού. Σας ευχαριστώ. Grazie, la parola di nuovo a Mr. Ο κ. Διαμαντούρος έχει το λόγο για να ανταπαντήσει. Και μετά θα αρχίσουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Grazie di nuovo. Euh, Κυρία Γκρουνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι πάντα δύσκολο να απαντήσει κανείς σε μια ερώτηση τύπου μήπως κάνετε υπερβολικά πολλά. Δεν θα ήμουν υποψήφιος αν ε, είχα την εντύπωση ότι η θητεία αυτή θα ήταν μία ε, θητεία υπερβολικά, υπερβολική, δηλαδή μετά από την εξαετή μου θητεία. Νομίζω ότι προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κάτι ως ε, διαμεσολαβητής προσπαθώ να χτίσω μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Πρόκειται για μια ε, μακρά και επίπονη διαδικασία. Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου κάνει την τιμή να με επανεκλέξει δια, διαμεσολαβητή, θα εμβαθύνω αυτά που ήδη έχω κάνει. Εσείς με ρωτήσατε κατά πόσο θα προσέβλεπα σε κάτι άλλο. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Ε, στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης των πολιτών και της πληροφόρησης έχουμε να κάνουμε με έναν ε, μεγαλεπίβολο στόχο ο οποίος απαιτεί πολλές προσπάθειες και εγώ είμαι έτοιμος να το προσπαθήσω, βάση περιπτώσει. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης ενός στόχου. Οι μεγάλοι άξονες δεν μπορούν να έχουν μεγάλη ευρύτητα, γιατί πάντα με απασχολούν θέματα κακοδιοίκησης, διαφάνειας, καταπολέμησης των κακοδιοίκησεων, έτσι ώστε να προσεγγίσω αυτό το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο σωστά. Για να απαντήσω σε μια άλλη σας ερώτηση, θεωρώ ότι η συνεργασία που προώθησα με την Επιτροπή Αναφορών διαχρονικά ήταν πολύ επικερδής και σημαντική για όλους. Ήδη προανέφερα ότι η επικύρωση συνθήκης της Λισαβόνας και η θέση της ισχύ από αύριο το πρωί είναι ύψης της σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Διανοίγονται πολλές δυνατότητες έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια. Και επειδή εγώ ήδη διαθέτω ένα δίκτυο συνεργασίας με συνηγόρους του πολίτη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μπορώ να συνεργαστώ για θέματα καλής ή κακής διοίκησης έτσι ώστε να δράτω με τις ευκαιρίες κάθε φορά που μου παρουσιάζεται για να προωθήσω κάτι περισσότερο. Αλλά θα με βοηθήσει πάντα η υποστήριξη της Επιτροπής Αναφορών, υποστήριξη την οποία πάντα είχα μέχρι τούδε. Βεβαίως, το θέμα συνεργασίας με τους άλλους φορείς ή με τους άλλους γενικότερα Εάν πρόκειται για τους εθνικούς ε, διαμεσολαβητές και τους περιφερειακούς ε, συνηγόρους ε, του πολίτη, θα χρησιμοποιήσω τη συνθήκη της Λισαβόνας για να ενισχύσω το δίκτυο του, των διαμεσολαβητών των κρατών μελών για να προχωρήσω πιο μακριά από ό,τι καταφέραμε μέχρι του παρόντος. Αυτό το οποίο είναι φοβερό και ελπιδοφόρο είναι ότι δεν υπάρχουν ποτέ όρια. Πάντα μπορούμε να ε, φευρίσκουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάτι το οποίο με παθιάζει εμένα προσωπικά και οι συνάδελφοι σε εθνικό επίπεδο πάντα αντιδρούσαν ενθουσιοδός ως προς τη δυνατότητα μεγαλύτερης συνεργασίας. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης σχέσεων και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση αν επανεκλεγώ. Ε, Κύριε Μποστινάρη, να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας. Για τον κοινό μηχανισμό. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι εγώ ως ε, διαμεσολαβητής και ο προκατοχός μου έχουμε επωφεληθεί πολύ από την προθυμία της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου σας να υποστηρίξει τη δράση μας. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί το σημείο κίνησης. Με άλλα λόγια, η ενίσχυση της περαιτέρω συνεργασίας, προκειμένου να μην κολλάμε στα ίδια, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί πραγματικά εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη στο σημείο αυτό. Ο διαμεσολαβητής ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργαστεί σε πολλαπλά επίπεδα με τους εθνικούς και περιφερειακούς ε, συνηγόρους και διαμεσολαβητές. Έχουμε αναπτύξει ήδη ένα σύστημα όπου οι εθνικοί περιφερειακοί διαμεσολαβητές υποβάλλουν ερωτήματα προς τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για διευκρινήσει, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και τώρα θα ήθελα να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η συνεργασία, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας θα ανοίξει και την δυνατότητα διακοινοβουλευτικών επαφών. Δηλαδή, εγώ θα μπορώ να ενθαρρύνω τους εθνικούς ομολόγους μου να έχουν επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια και έτσι αυτό το δίκτυο, αν θέλετε, να καταστεί πολύ πιο ζωντανό. Και έτσι, στην πορεία, να τραβήξουμε και την προσοχή των πολιτών πέρα από το θέμα των ετοιμάτων αυτών που υποβάλλονται προς το διαμεσολαβητή, έχουμε χρησιμοποιήσει την ήδη υφιστάμενη δομή του δικτύου. Έχουμε ένα φόρουμ συζήτησης και το οποίο και χρησιμοποιούμε για να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συναδέλφους σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του θεσμού του διαμεσολαβητή για θέματα υγείας, σε ό,τι αφορά δηλαδή τους ασθενείς. Κάποιοι ανησυχούν όταν ακούν ότι υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά μέσα από το φόρουμ, μέσα από το δίκτυο ήρθαν και απευθύνθηκαν σε μας, διευκρινίσαμε το θέμα και καταφέραμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνεργασίες, συνέργειες, προκειμένου και να επιληθεί το ζήτημα, αλλά και να βοηθήσουμε τους θεσμικούς, ε, τις θεσμικά όργανα να κατανοήσουν τις ανησυχίες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λοιπόν ανάγκη να υπάρξει απαραίτητα ένας κοινό μηχανισμός. Θα ήθελα μάλλον να ενισχυθούν οι ήδη υφιστάμενοι μηχανισμοί, να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου να υπάρχει μια στρατηγική πολλαπλών επαφών συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Διαμεσολαβητή, των άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου, των εθνικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες που τελικά θα έχουν αποτέλεσμα για τον πολίτη. Κύριε Χάνκη, να σα ευχαριστήσω για την ερώτηση που μου κάνατε. Ξέρω από πού προέρχονται οι ανησυχίες σας. Ξέρω ότι στη χώρα σας έχετε διαμεσολαβητή για τις μειονότητες. Συνεργάστηκα με τον κύριο Κάλτενμπαχ όσο διατέλεσε διαμεσολαβητής για τις μειονότητες και ξέρω ότι δυστυχώς το θέμα των μειονοτήτων αποτέλεσε πολύ σημαντικό θέμα στην όλη ιστορία της περιφερειάς σας. Το γνωρίζω λοιπόν και ως διαμεσολαβητής, αν επανεκλεχθώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό. Να σας πω ότι και το γνωρίζω το θέμα και με απασχολεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να διευκρινίσω και άλλα δύο στοιχεία. Προφανώς, ως Ευρωπαίος διαμεσολαβητής έχω λάβει εξαιρετικά μικρό αριθμό καταγγελιών σε ό,τι αφορά τις μειονότητες. Οι πιο πολλές καταγγελίες που λαμβάνω έχουν να κάνουν με παραβιάσει των, δικαιώμα, των δικαιωμάτων των Ρωμά στα κράτη-μέλη και ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο είναι ότι όλα αυτά τα θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου, γιατί εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συναδέλφων μου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αλλά αν κατανοήσουμε, αν ερμηνεύσουμε τις μειονότητες υπό την ευρύτερη έννοια, οι ευάλωτες ομάδες δεν είναι μόνο εθνοτικές μειονότητες. Αν λοιπόν το ερμηνεύσουμε έτσι, προφανώς ο διαμεσολαβητής έχει πεδίο αρμοδιότητας σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διακριτική μεταχείριση βασιλικίας. Έλαβα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα και αν θέλετε βαρύνουσας ηθικής σημασίας υπέβαλα και ειδική έκθεση προς την Επιτροπή σας και προς το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης ξεκίνησα μια έρευνα πρωτοβουλίας και μια δημόσια διαβούλευση για τα ευάλωτα άτομα σε ό,τι αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήταν πολύ ευρύ το πεδίο αυτό. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχω αναλάβει πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και αυτό καταδεικνύει ότι ο διαμεσολαβητής έχει ήδη αναλάβει δράση σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες, εντός φυσικά πάντα της αρμοδιότητάς μου. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, είμαι έτοιμος, είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, με το Ευρωκοινοβούλιο, με την Επιτροπή, με τους συναδέλφους μου σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο, για να καταργήσω αυτή τη δομή των διπλών μέτρων στην οποία αναφερθήκατε. Πάντα φυσικά εντός των περιορισμών που μου επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Κύριε Διαμαντούρο, θα ήθελα να, είσαστε, να συγκεφαλαιώσετε περισσότερο και δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία ΚΑΣΤΕΑΗ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα είναι το πρόβλημα, αυτό το συνηθισμένο πρόβλημα. Προσπαθούμε να είμαστε συνοπτικοί και να αναφέρουμε τα πάντα, αλλά τελικά δεν έχουμε χρόνο, κυρία Γκούντς, Μιλήσατε για την μείωση του αριθμού των καταγγελιών. Ασφαλώς και μείωση των αριθμών των καταγγελιών και, όπως σας είπα, τρει μήνες ε, παίρνει η αντιμετώπιση της πιο απλής καταγγελίας. Και να μην ξεχνάτε ότι έχω και 23 γλώσσες πάντα να λάβω υπόψη μου. Προσπαθώ λοιπόν να μειώσω το χρόνο απάντησης ε, των, στις καταγγελίες των πολιτών και ελπίζω να το πετύχω. Κυρία Γουάλης, σας ευχαριστώ και βρίσκομαι υποχρονική πίεση. Το θέμα της κοινή πύλης. Ασφαλώς κυκνηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού οδηγού που δημιουργήθηκε στην αρχή του έτους στα πλαίσια της ιστοσελίδας μας. Μέσω αυτού του οδηγού λοιπόν, ο πολίτης μέσω απαντήσεων και ερωτήσεων θα μπορέσει να κατευθυνθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα ναι, αυτή η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινούμαστε. Συμμετέχουμε και στην διαδικασία, αν θέλετε, απάντησης τηλεφωνημάτων. Αν θέλει δηλαδή ο πολίτης μπορεί να λάβει άμεση απάντηση, χωρίς καθυστέρηση. Σε ό,τι αφορά τη Λισαβόνα και το Συμβούλιο και την διαφάνεια, ξέρετε ότι έχω υποβάλει προς το Κοινοβούλιο μια ειδική έκθεση η οποία είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια στο Συμβούλιο και ανυπομονώ ασφαλώς να συνεργαστώ και με το νέο Συμβούλιο εφόσον επανεκλεχθώ και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τις νέες δυνατότητες της συνθήκης της Λισαβόνας αλλά το Κοινοβούλιο αυτό θα έχει νέες δυνατότητες να συνεργαστεί με πιο μεγάλη διαφάνεια με το Συμβούλιο επίσης και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τη δυνατότητα συνεργασίας που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας για συνεργασία λοιπόν με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρία Άουκεν. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σας, αλλά δεν είναι εύκολο να τις απαντήσω γρήγορα. Να σας πω ότι το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση για την εφαρμογή του νόμου σε ό,τι αφορά περιπτώσεις καλής διαχείρισης. Και είμαι φυσικά πρόθυμος να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής σας και του Διαμεσολαβητή για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πολίτη. Αλλά ασφαλώς αυτό αποτελεί τμήμα, αν θέλετε, μιας νομοθετικής δράσης, την οποία θα ήθελα να συνδράμω για το πώς μπορούμε να ε, κάνουμε καλύτερη εποπτεία, παρακολούθηση, νομίζω μέσω της εντατικοποίησης των δράσεων του διαμεσολαβητή. Και αυτό προσπάθησα να σας ε, περιγράψω. Αν επανεκλεχθώ, σκοπεύω να στραφώ όλο και περισσότερο προς τα θεσμικά όργανα και συγκεκριμένα προς τις υπηρεσίες, προκειμένου αυτή η κουλτούρα της εξυπηρέτησης του πολίτη τελικά όντω να αποβεί προς όφελο του πολίτη. Κύριε Τσίζεστερ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Η καλύτερη απόφαση που έλαβα. Μου φαίνεται ότι μία από τις καλύτερες αποφάσεις μου, για να μην σας πω η κατεξοχή είναι καλύτερη απόφασή μου, ήταν η ειδική έκθεση που υπέβαλα στο Κοινοβούλιο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ήταν μια στιγμή κατά την οποία μπόρεσα να ασχοληθώ με μια βασική ανησυχία σε κοινωνικό επίπεδο. Παιδιά, ειδικέ ανάγκες, ειδική εκπαίδευση είναι σημαντικά θέματα στην ε, νομική τάξη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μετανιώνω. Θα σας δώσω την απάντηση ότι θα σας δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να αποφύγω να απαντήσω. Πάνω από μία απόφαση έχω μετανιώσει. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρουσιάσω σαφώς τις θέσεις μου στο Κοινοβούλιο σε θέματα που είχαν να κάνουν ε, με τους, τις αποζημιώσεις των, ε, των βουλευτών, παρότι καταλήξαμε σε πολύ καλό αποτέλεσμα. Απέτυχα όμως να εξηγήσω σαφώς το θέμα αυτό. Αυτό θα ήθελα να το είχα κάνει διαφορετικά. Πώς να θεσμοποιήσουμε την παρακολούθηση. Νομίζω ότι σας έχω εξηγήσει αρκετά πώς μπορώ. Πώς θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να μπορώ να χρησιμοποιήσω το προσωπικό μου, όχι μόνο εμένα, για να θεσπίσω επαφές ε, με την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω ελληνικά τώρα. Είμαστε υπό ασφιχτική πίεση. Ho già detto che c'è Νομίζω ότι ήδη σας απάντησα για το πώς προτίθεμαι να συνεργαστώ με τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, ε, άρα επιτρέψτε μου να μην το αναπτύξω. Ε, το θέμα της ε, προαγωγής ενός ε, πνεύματος εξυπηρέτησης ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχω ήδη αναπτύξει και το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί βασικά με την εντατικοποίηση των επαφών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με τους θεσμούς. Το ότι οι θεσμοί αυτοί δεν είναι εκλόγιμοι δεν μειώνει την ευκαιρία που μου παρέχεται να μπορέσω συστηματικά να συζητάω με το Κολέγιο των Επιτρόπων, με τους Επιτρόπους, με τους Γενικούς Διευθυντές και επίσης με τους άλλους μεγάλους θεσμούς. Το πώς η ε, πολίτες θα μάθουν περισσότερο για τα δικαιώματά τους. Αυτό νομίζω περνάει οπωσδήποτε μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η Λισαβόνα και μέσα από τα εθνικά κοινοβούλια. Για μένα τα εθνικά κοινοβούλια είναι κρίσιμος μηχανισμός προσέγγισης. Κύριε Σαλαβράκο, τελευταία ερώτηση. νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει και απλώς να τονίσω ότι και πάλι ότι για μένα η Λισαβόνα ανοίγει πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τις οποίες θα ήθελα να αξιοποιήσω εφόσον μου δοθεί η τιμή μιας νέας εκλογής. Ευχαριστούμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα και θέλω να σας συγχαρώ και για κάτι ακόμη. Για την πληρότητα των απαντήσεών σας, αλλά κυρίως για την ειλικρίνεια που διέκρινε τις απαντήσεις σας. Ε, δύο πράγματα μόνο Απαντώντας στην ερώτηση για το τι θα πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερες ε, υπηρεσίες στους Ευρωπαίους πολίτες, επισημαίνεται έξι σημεία, ανάμεσα από τα οποία εγώ ξεχωρίζω δύο. Το πρώτο είναι η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών. Και το δεύτερο είναι η παροχή εξηγήσεων για το έργο τους, σε γλώσσα κατανοητή για τους πολίτες. Είναι δύο σημεία καθοριστικά κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί μέσα από τη δική σας δουλειά μπορεί να προαχθεί κατά αποτελεσματικό τρόπο αυτό που συνηθίζουμε να λέμε γενικά, αλλά που έχει ιδιαίτερο ειδικό ενδιαφέρον, η ευρωπαϊκή ιδέα. Και επειδή ε, βλέποντας τα πεπραγμένο σας και ακούγοντας τις τεκμηριωμένες και ειλικρινείς, επαναλαμβάνω, απαντήσεις σας, ε, περιμένω πάρα πολλά από σας και ελπίζω. Να, να δηλώσω ε, και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους εδώ της Επιτροπής ότι με την περίπτωση της εισήγησης για την έκθεση του κυρίου Διαμαντούρου για το 2008 ε, εξάντλησα τα όρια της αντικειμενικότητάς μου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι είχα την εξαιρετική τιμή να λειτουργήσω όχι ως Ελληνίδα πέραν της έναν Έλληνα, αλλά ως ένα μέλος ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλαβα την υποχρέωση να εισηγηθώ για ένα άλλο όργανο θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εντελώς συμπτωματικά έτυχε να είναι Έλληνας και για το οποίο πραγματικά τώρα μπορώ να σας πω πόσο καμαρώνω που ε, ανέλαβα αυτή την τεράστια ευθύνη. Θα τελειώσω με μία ερώτηση κύριε Διαμαντούρα. Μιλήσατε κάπου και διαβάσαμε και, στις, ε, και στην έκθεσή σας για τις αυτεπάγγελτες έρευνες. Σε ποιους τομείς θέλετε να μας πείτε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Ράπτη και την κυρία Παλιαδέλη για τα καλά τους λόγια. Ευτυχώς επειδή δεν έχει πολύ φως δεν φαίνεται πόσο έχω ερυθριάσει με τα υπερβολικές, υπερβολικές φιλοφρονήσεις. Αλλά τις ευχαριστώ παρά τα αυτά. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ράπτη, ε, να πω ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι είναι απέτηση ενός από έναν όμπουτσμαν να είναι ειλικρινής. Και άρα εκείνο το οποίο κάνω είναι προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες του θεσμού, όντας ειλικρινής, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά την απλή γλώσσα, θεωρώ ότι και πάλι ο Ombudsman έχει τον, ε, την υποχρέωση να μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες σε γλώσσα η οποία είναι κατανοητή. Και γι' αυτό έχω επιχειρήσει και έχω απλοποιήσει και τη γλώσσα των αποφάσεών μου και τη ετήσια έκθεση και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και το έχω και εσωτερικά στο θεσμό εφαρμόσει και ευελπιστώ να το εφαρμόσω ακόμα περισσότερο εάν μου δοθεί η ευκαιρία να το κάνω. Σας ευχαριστώ για αυτές τις δύο παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά τέλος την κυρία Παλιαδέλη, κοιτάξτε, οι αυτεπάγγελτες έρευνες είναι ένας πάρα πολύ, σημαντικός, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον διαμεσολαβητή. Πρέπει να χρησιμοποιείται λοιπόν με φιδό και πρέπει να χρησιμοποιείται για κέρυε ευκαιρίες. Οι κύριες ευκαιρίες μπορεί να είναι είτε αυτό που λέμε συστημική κακοδιοίκηση, δηλαδή πολλά φαινόμενα σε ένα θεσμό το οποίο μας οδηγούν να το κοιτάξουμε, είτε παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος έστω και από ένα άτομο. Με αυτόν τον τρόπο έχω λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια και αυτόν τον τρόπο ε, προτίθεμαι να λειτουργήσω και στο μέλλον. Δηλαδή να κάνω χρήση της αυτοπάγγελης έρευνας προκειμένου να αναδείξω προβλήματα συστημικά και να βοηθήσω να, αν θέλετε, να διαπαιδαγωγήσω τους θεσμούς πάλι προς την κατεύθυνση της έννοιας του πνεύματος και του πολιτισμού εξυπηρέτησης προς τους πολίτες. Ε, Υπάρχει ένα αίτημα ε, Χάρκιν εκτός χρόνου. Έχουμε δύο λεπτά ή δυνατόν σας δίνω το λόγο, ένα λεπτό σε εσά και ένα λεπτό στον κύριο Διαμαντούρο για να απαντήσει. Χάρκιν. Εντάχει. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήμουν ε, εξ αρχής της ακρόασης. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας τιμώ, αλλά έπρεπε να βρίσκομαι αλλού. Πρέπει πολλές φορές να είμαστε πανταχού παρόντες. Θίξατε το θέμα των εξόδων των βουλευτών και έχει μεγάλη ε, σημασία γιατί δεν μπορούμε να, το, ε, να αναφερθούμε σε αυτό αλλού. Μιλήσατε για το κατά πόσο πρέπει να είναι κανείς κατανοητός σε μία γλώσσα. Όχι πάντα στη μητρική γλώσσα όλων, αλλά οι πολίτες δεν ξέρουν πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα πάντα. Τελείωσε το λεπτό μου. Ε, ξέρω ότι διανύσατε μία απόσταση, έχετε περαιτέρω σχέδια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες κατανοούν τις απαντήσεις και ότι σε αυτές τις απαντήσεις δεν υποσχόμαστε στους πολίτες περισσότερο από αυτό που μπορούμε να τους δώσουμε. Εκτιμώ το σχόλιο σας και είμαι ευγνώμων για το ότι αναγνωρίσετε το θέμα των επιδομάτων των βουλευτών που έθιξα. Ως προς το ερώτημά σας κάθε αυτό, θα σας το θέσω ως εξής. Το εκπληκτικό θέμα της καλοδιαχείρισης είναι ότι είναι ανοιχτό. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενεργητικοί. Ε, άρα γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν πρέπει να υπερβώ ορισμένα όρια, αλλά πρέπει να είμαι ε, ιδιαίτερα ενεργητικός και να διαδραματίσω ενεργό ρόλο σε αυτό το τομέα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου είπατε ότι θα πρέπει να εξισορροπήσω, να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες και χαμηλές αποδόσεις. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Προσπαθώ να υπόσχομαι λίγα και να παρέχω πολλά εκεί που μπορώ. Και έτσι προσπαθώ να κινηθώ. Αλλά εκτιμώ τα σχόλιά σας και προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω απλή γλώσσα Βεβαίως η ουρανή είναι το όριό μας πάντα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας και να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι και ενεργητικοί. Ευχαριστούμε κύριε Διαμαντούρο. Να σας χαιρετήσουμε και να περάσουμε στον τελευταίο υποψήφιο. Ο κύριος Place Mrs. Mazzoni. Ε, να καλώσουμε τον κύριο ε, Μονέ, να του δώσουμε χρόνο να εγκατασταθεί. For the next 15 minutes. Μπορείτε να μας κάνετε την ε, εισήγησή σας για τα επόμενα 15 λεπτά.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 Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να υποβάλω την υποψηφιότητά μου ενώπιον της Επιτροπής σας. Θα κάνω την παρουσίασή μου σε τρεις γλώσσες. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανανέωση, ο ανανεωτισμός. Δηλαδή, βλέπουμε νέα, με καινούρια μάτια, τον ρόλο του Ευρωπαίου Ομπουτσμαν και θέλω να δώσω ε, απαντήσεις στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι ότι είμαι επαγγελματίας του τομέα. Ήμουν όπως ξέρετε, ομοσπονδιακός ομπουτσμαν στην χώρα μου, στο Βέλγιο, από το 1997 μέχρι το 2005. Τώρα είμαι καθηγητής στην Μπρουζ στο, στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό και προβάλλω έναν εναλλακτικό τρόπο ε, επίλυσης των διαφορών. Επίσης είμαι νομομαθής αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να προωθήσω το ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή και αυτό το κάνω και ως νομομαθής. Δηλαδή το δίκαιο πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο για μένα είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο για να γίνει κανείς διαμεσολαβητής, διότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό να είναι κανείς νομομοθής για να προβάλλει υποψηφιότητα συνηγόρου του πολίτη. Επίσης γνωρίζω τα ευρωπαϊκά όργανα και τους θεσμούς, καθώς και τα ευρωπαϊκά γραφεία στο Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, ε, Κοπενχάγη, μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Συνεργασίας και έχω δημοσιεύσει άρθρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία της. Ένα άλλο ε, ατού, ας το πω έτσι, είναι ότι ομιλώ πέντε ευρωπαϊκές ε, γλώσσες και πιστεύω ότι έχει σημασία να σεβόμαστε την ταυτότητα του καθενός και τη γλώσσα του που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς του και αυτό που έχει, ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Η τελευταία πτυχή της υποψηφιότητάς μου είναι ότι πρόκειται για μία ε, διαγενειακή, ας το πω έτσι, υποψηφιότητα. Είμαι 49 χρονών, μεταξύ δύο γενεών δηλαδή, και μπορώ να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις και να εργαστώ για να επιλύσω ε, σημαντικά ζητήματα. Πρόκειται για μια ηλικία μεταξύ δύο γενεών δηλαδή. Και πιστεύω ότι μπορώ να επιλύσω πολλά χάσματα. Θεωρώ για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ότι θα πρέπει να διδραματίσει σημαντικούς ρόλους σε ό,τι αφορά τους στόχους της ενίσχυσης της δημοκρατικής εποπτείας στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσω της, του ρόλου κλειδί, αν θέλετε, του διαμεσολαβητή, επιτυγχάνεται και καλύτερος έλεγχος σε εθνικό επίπεδο και ως κοινοβουλευτικός ε, διαμεσολαβητής σημαντικό είναι να συνδράμει κανείς στα εθνικά κοινοβούλια για τον εκδροματισμό της ε, Ένωσης. Το κοινοβούλιο είναι το όργανο με την <laughs> μεγαλύτερη νομιμοποίηση στο ιστορικό των της Ένωσης. για να προσδώσει και αυτό το χαρακτήρα στα ευρωπαϊκά θεσμορπα... θεσμικά όργανα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να εισέλθουν στον πυρήνα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς η αρχή της διαφάνειας θα πρέπει να καταστεί η διαφάνεια χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 1 της συνθήκης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια σε, όλες τις, ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα, σε όλες τις υπηρεσίες της Ένωσης και θα πρέπει λοιπόν να καταστεί προτεραιότητα υπαριθμών 1 για τον διαμεσολαβητή. Η λογοδοσία επίσης αποτελεί το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο από τις βασικές αυτές αρχές σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η τρίτη αρχή, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι ο πολιτισμός της εξυπηρέτησης. Αυτή λοιπόν η αρχή θα πρέπει να αποτελεί μια θεμελιώδη προϋπόθεση και θα πρέπει να τεθεί στον πυρήνα των υπηρεσιών και θα πρέπει να αποτελεί την τροπία του κάθε υπαλλήλου της Ένωσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει ένας άλλος στόχος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να είναι η ενίσχυση των θεμελιδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την χάρτα των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, αναπήρων, σε ό,τι αφορά ζητήματα αλληλεγγύησης και το καθεξής. Αυτά πιστεύω είναι θεμελιώδη ζητήματα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποτελεί πηγή μεταρρυθμίσεων να προτείνει μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. για να τεθεί, αν θέλετε, η διαδικασία μεταρρύθμισης αυτή πιο πολύ στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του πολίτη. Και μεταρρύθμιση για να τύχουν αναγνώρισης οι αρχές καλής διαχείρισης και να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σκληρή δουλειά για να πετύχω τους στόχους που ανέφερα ως Άνω, θεωρώ ότι θα μπορούσα να βοηθήσω προκειμένου να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να αυξηθεί και η ευαισθητοποίηση του Ευρωπαίου υπαλλήλου για το ρόλο που διδραματίζει ως βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνουν δράσεις για να βελτιωθεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Και τώρα θα περάσω στις συγκεκριμένες προτάσεις που θέλω να προτείνω. Καταρχάς, ε, οι συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις θα εστιαστούν στην καλύτερη ευρωπαϊκή διαχείριση. Καταρχάς, για να εποπτεύεται η πλήρης εφαρμογή της καλής διοικητικής συμπεριφοράς, όχι μόνο από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα, αλλά από όλες τις υπηρεσίες της Ένωσης, ειδικά μετά από τη σχετική απόφαση τον Οκτώβριο του 2008. Ένα άλλο στοιχείο θα ήταν η ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα καλής ε, διοικητικής συμπεριφοράς. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι θα χρειαζόταν ε, διαθεσμικός διάλογος που θα εμπλέξει όλες τις υπηρεσίες, όλα τα θεσμικά όργανα. Και επίσης θα ήθελα να οριστεί καλύτερα ο όρος της κακοδιαχείρισης για να συμπεριληφθούν πιο πολλές ε, πτυχές από τη σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να διοριστεί και ένας ε, υπεύθυνο για τη διαφάνεια σε κάθε, ξεχωριστά σε κάθε ευρωπαϊκό όργανο και υπάρχει και μια εξαιρετική σχετική έκθεση του κυρίου Κάσμαν. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται η θέση αυτή. Τέλος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να, να παρακολουθεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και φυσικά να πάει πολύ παραπέρα από την εφαρμογή αυτή. Κατά δεύτερον, η ανάγκη να, να αυξηθεί η σημασία και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Υπήρξε αύξηση των καταγγελιών μεταξύ 2003 και 2008 κατά 28,5%. Να δούμε πόσες από αυτές τις καταγγελίες ήταν παραδεκτές. Η αντίστοιχη αύξηση ήταν 15% και κατά κεφαλή η αύξηση αυτή είναι λιγότερο από 1% επειδή οι καταγγελίες, οι έρευνες, ε, μάλλον τελικά η αύξηση, η μείωση των ε, ερευνών ήταν 16,3%. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφημίζουμε πιο πολύ τα δικαιώματα των πολιτών να αναφέρονται και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη συνεργασία με τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επαφή με τους πολίτες και θα ήθελα συνεχή συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια να δημιουργηθεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο απεσταλμένων του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τη μόνιμη την προσωπία της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής με τα διάφορα κέντρα ενημέρωση στα κράτη-μέλη που υφίστανται ήδη και τέλος θα ήθελα να προτείνω οι διοικητικές αποφάσεις να αναφέρουν το δικαίωμα του πολίτη να προσφεύγει στον διαμεσολαβητή. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μαζί με καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών όταν ε, κάνουν καταγγελίες. Και θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα προκαταρτικών ερωτήσεων. Θα πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των μη παραδεκτών καταγγελιών, γιατί σήμερα ανέρχονται σε 85% του συνόλου των καταγγελιών και αυτό μας εμποδίζει στο έργο μας και θα ήθελα να δημιουργηθεί ένας διατραστικός οδηγός, ο οποίος θα είναι ίδιος για όλα τα θεσμικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις σχετικές ιστοσελίδες. Μία τρίτη σειρά δράσεων θα εστιαζόταν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό. Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των ε, Ευρωβουλευτών. Ξέρετε ότι το λιγότερο από 10% των καταγγελιών έχουν υποβληθεί από ευρωβουλευτές. Σε ό,τι αφορά δηλαδή καταγγελίες οι οποίες προέρχονται από την εκλογική περιφέρεια του κάθε βουλευτή. Αυτό καταδεικνύει ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να βρει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για να υποβάλλονται τέτοιες καταγγελίες. Συνεργασία μεταξύ του διαμεσολαβητή και της Επιτροπής σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε η συνεργασία ήταν πάντα εξαιρετική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών και επίσης μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και άλλων επιτροπών, μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των εθνικών ή περιφερειακών συνηγόρων και των σχετικών επιτροπών αναφοράς. Λειτουργεί το σύστημα, όχι όμως επαρκόξ. Το 2008 μόνο 8 νόμοι ξεκίνησαν από τέτοιες κοινέ δράσεις. 8 μόνο δεν αρκούν φυσικά αυτοί οι αριθμοί. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνέργειες στο δίκτυο αυτό. Ζητώ επίσης μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητή και των Εθνικών Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εφαρμοστεί ο δοσμευτικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέλος μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για περιπτώσεις συνεχούς και επανελειμμένης κακοδιαχείρισης, όπου έχουν ε, εκδοθεί συστάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τέταρτη και τελευταία σειρά δράσεων και προτάσεων έχει να κάνει με τη βελτίωση των δράσεων του ίδιου του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει την σωστή χρήση του άρθρου 226 και 228 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση, όπως τα γνωρίζετε. Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο της ε, καλύτερης ε, ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της οποίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και διαδικαστικά θέματα, αλλά και θέματα επί της ουσίας. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η διάρκεια των ερευνών. Έχει ήδη βελτιωθεί κατά μέσο όρο 13 μήνες διαρκεί μία έρευνα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση των κρίσιμων παρατηρήσεων, των ε, κριτικών που γίνονται προκειμένου να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα εθνικά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε περιπτώσει κακοδιαχείρισης. Και τέλος, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει την πιο απλοποιημένη διαδικασία, πιο απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης και τις πιο απλοποιημένες λύσεις για την εξέβρεση συνένεσης. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφόρων. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αν έχετε ερωτήσει, είμαι στη διάθεσή σας. Ε, Ξεκινάει η συζήτηση. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Μονέ μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το, την επόμενη θητεία του Ευρωπαίου ε, Διαμεσολαβήτη. Ποιες είναι οι βελτιώσεις που προβλέπετε για το ρόλο του Διαμεσολαβήτη και εάν πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός, η θέση του Διαμεσολαβήτη. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη συγκεκριμένη ευθύνη του διαμεσολαβητή όπως ορίζεται από τις συνθήκες και χωρίς να μιλήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα, ποια είναι τα χάσματα ή τα κενά που διαβλέπετε στη θέση αυτή μέχρι τώρα. Πώς θα θέσετε σε εφαρμογή το σχέδιό σας, γιατί ίσως είναι δύσκολο να ε, καταφέρει κανείς τα πάντα πώς θα συνεργαστείτε με την Επιτροπή Αναφορών, αν μπορείτε να μας μιλήσετε συγκεκριμένα και πώς προβλέπετε τη συνεργασία σας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μποσινάρου. Ευχαριστώ. Κύριε Μονέ, η Επιτροπή Πέτη με ανησυχία ανέφερε ότι το 2008 ότι το 36% των προσφυγών σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη ε, πληροφόρησης ή μη χορήγηση πληροφοριών και εγγράφων. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό έτσι ώστε να ε, οικοδομήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ποια είναι η πρότασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άγκης. Ε, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Μονέτ, θα ήθελα να σας υποβάλω μία σειρά σύντομων ερωτήσεων που σχετίζονται με όλα όσα μας παρουσιάσατε ανάμεσα στους στόχους σας, δηλαδή η βελτίωση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ύψης της σημασίας, διότι εργαζόμαστε για τον Ευρωπαίο πολίτη και όχι το αντίστροφο. Η πρώτη μου ερώτηση έχει ως εξής. Ποιες εγγυήσει μπορείτε να μας παράσχετε έτσι ώστε να μην υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων. έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ισότητα δικαιωμάτων όλων των προσφευγόντων. Να μην υπάρχει πολίτης δεύτερης κατηγορίας για γεωγραφικούς λόγους ή για τη χώρα στην οποία ανήκει. Μιλήσατε στην αρχή της παρέμβασής σας για μία νέα ε, όθηση, όθηση σε σχέση με το χάσμα των γενεών θα μελετήσετε όλες τις ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, υποψίες διαφθοράς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για, τις υψηλότερα, για τα υψηλότερα κλιμάκια ενός κρατικού μηχανισμού. Όταν μιλάμε μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με αντικρουόμενες, όχι αντικρουόμενες, αλλά θέσεις που βρίσκονται η μία στον αντίποδα της άλλης. Μιλάμε για καταπολέμηση τρομοκρατίας, για οργανωμένο έγκλημα και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να υπερβούμε ε, με ορισμένες οριοθετήσεις που έχουν γίνει. Θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς το συσχετισμό μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Επίσης και μία άλλη ερώτηση. Με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούν να υπάρξουν και άλλες αναφορές σε σχέση με δημοψηφίσματα. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων μειονοτήτων που είναι συλλογικά δικαιώματα, όπως γίνεται τώρα στη Σλοβακία, όπου υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων της ε, ουγγρικής ε, μειονότητας. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά, γιατί η ουγγρική μειονότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική της ε, γλώσσα. Κύριε Παλιαδέλη. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική παρουσίαση ε, όσων πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν προκειμένου ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής να ανταποκριθεί στο όραμα που έχετε εσείς δημιουργήσει για αυτόν. Μία πολύ απλή ερώτηση. Πώς σκέφτεστε να μειώσετε τη διάρκεια των ευρωπαϊκών των, των ερευνών που, που έχουν σχέση με τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή. Reduce the duration of the uh, European Ombudsman inquiries. Practically, meaning. Ευχαριστώ. Χάρκιν, ευχαριστώ πρόεδρε. Και καλησπέρα σας κύριε Μονέτ. Σας ευχαριστούμε για την ε, πολύ εμπεριστατωμένη και πρακτική παρουσίαση που μας κάνατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Σύντομες. Και θα ήθελα κυρίως να σας ζητήσω να μας δώσετε παραδείγματα για τα θέματα που δείξατε στην παρουσίασή σας. Μιλήσατε για το πώς θα περάσουμε από τα κλασικά νομικά ένομα δικαιώματα στις ένομες νομικές προκλήσεις. Τι ακριβώς εννοείτε. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα. Επίσης αναφέρατε στην επιχειρηματολογία σας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του υπηρετικού, του ευρωπαϊκού και του αγγλοσαξονικού συστήματος, νομικού συστήματος και ότι υπάρχει ανάγκη φυσικά να γίνουν και τα δύο σεβαστά, αν θα θέλετε να αναπτύξετε το θέμα αυτό. Επίσης είπατε ότι ο νόμος πάντα θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Έχετε κάτι συγκεκριμένο υπόψη σας, κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούν καλύτερα να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του πολίτη. Τέταρτη ερώτηση. Μιλήσατε για κακοδιαχείριση και ότι θέλετε να διευρυνθεί ο ορισμός αυτός. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε, αν θα μπορούσατε να επαναλάβετε παρακαλώ. Και τέλος, μιλήσατε για την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών σε ό,τι αφορά την ε, διερεύνηση των ίδιων θεμάτων. Έχετε κάτι συγκεκριμένο υπόψη σαν σας, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πολλά υπόσχονται αυτά που μας είπατε. Είπατε ότι θα βελτιώσετε την παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάση και το είπατε αυτό και όσον αφορά τη διαδικασία και όσον αφορά το περιεχόμενο των δράσεων της Επιτροπής στον τομέα αυτών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περαιτέρω πώς θα παρακολουθείτε τις αποφάσεις της Κομισιόν επί της ουσίας. Και επίσης είπατε ότι ελάχιστες φορές, ίσως ποτέ, οι, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ε, ασκήσει το δικαίωμα τους να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πού σας λείπουμε, πού θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα τη δουλειά μας. Τι υποθέσεις θα έπρεπε να έχουμε υποβάλει στον διαμεσολαβητή, διότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας κατηγορείτε, μπορεί να έχετε πολύ σοβαρά πράγματα κατά νου που παραλείψαμε. Και είμαι πολύ περίεργη να ακούσω Πού δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Ο κύριος Σαλαβράκος. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ, σε μια ισορροπία σχέσεων Όμπουσμαν και Επιτροπής Αναφορών. Και θα παρακαλούσα να μου πείτε, εάν βλέπετε κάπου θεσμικά να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ποιες είναι κατά την άποψή σας που δημιουργούν μια δυσλειτουργία στην άσκηση των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του Όμπουσμαν. Ευχαριστώ. La parola di nuovo Mr. Monet. Um, a lot of questions, Mrs. President. Πολλές ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ξεχάσω καμία. Κυρία Γκρούνη, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Με ρωτήσατε Ποιε είναι οι προτεραιότητες Ποια είναι μάλλον η προτεραιότητα την οποία ξεχωρίζω μεταξύ των όσων ανέφερα. Πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω μία, γιατί φυσικά πολλά θέματα είναι κατεπίγοντα. Θεωρώ ότι αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω μία προτεραιότητα θα ήταν το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στον διαμεσολαβητή και νομίζω ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνεται σωστά και αυτό θα αποτελούσε την κορυφαία προτεραιότητά μας γιατί η θέση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή υπάρχει εδώ και 14 χρόνια και βλέπουμε όντως να αυξάνεται ο αριθμός των ε, καταγγελιών Κοιτώντας όμως τα αριθμητικά στοιχεία σε κάποιες ορισμένες χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση. Αλλά σε ό,τι αφορά το παραδεκτό των καταγγελιών, βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό. Γιατί δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αλλά στο πεδίο αρμοδιότητα του Εθνικού Διαμεσολαβητή. οι πολίτες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μια πολύ μικρή ομάδα. Μπορεί τελικά να καταλήξουμε να έχουμε εκατομμύρια προσφυγές αν είναι υπερβολικά ευρύς ο ορισμός, αλλά είναι μικρός αριθμός των ε, προσφυγών για τις οποίες είναι τελικά αρμόδιος ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή και ο προϋπολογισμός ε, του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή επικρίνεται σε πολλές περιπτώσεις από τους Ευρωπαίους, από τους Ευρωβουλευτές. Μπορεί να θεωρήσει κανείς δικαίως ε, εκ πρώτης όψεως ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για να αντιμετωπιστεί μεγάλος αριθμός μη παραδεκτών προσφυγών. Τουλάχιστον στο Βέλγιο επικρατεί αυτή η άποψη. Θα πρέπει λοιπόν για πολλούς και διάφορους λόγους να τονίσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με το δικαίωμά του να αναφέρεται και να προσφεύγει στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Ιδιαίτερα και με την ηλεκτρονική οδό, για να διασφαλίσουμε ότι τελικά οι καταγγελίες που καταλήγουν σε εμά είναι οι καταγγελίες επί των οποίων μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί το καταστατικό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουνα υπέρ της αναθεώρησης αυτής για συγκεκριμένους λόγους, τρεις συγκεκριμένους λόγους, αλλά Δύο εξ αυτών έχουν πλέον αλλάξει. Θα ήθελα λοιπόν οι αλλαγές αυτές να συμπεριληφθούν και να εφαρμοστούν. Και το άρθρο 4.3 επιτρέπει στον διαμεσολαβητή να ε, έχει πρόσβαση στα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του, στο, στην παράγραφο 9 του άρθρου 149 σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα απόρριτα έγγραφα. Πρόκειται για μια πολύ ωφέλιμη διάταξη η οποία δίνει εγγύηση στους ε, πολίτες ότι τα απόρριτα έγγραφα θα παραμείνουν απόρριτα. Αλλά όταν κάτι τέτοιο το λέει η δίκηση, υπάρχει πάντα η υποψία της μεροληψίας. Όχι όμως όταν προβαίνει σε τέτοιες αποφάσεις ο διαμεσολαβητής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχύεται η εμπιστοσύνη του πολίτη. Άλλο ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω παρακολούθησα τη σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάνθηκε ότι δεν επρόκειτο για θετική δράση σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, σε ό,τι αφορά την άμεση προσφυγή στο ΔΕΚ, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακοδιαχείριση. Νομίζω ότι δικαίως αποφάσισε, όπως αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωκοινοβούλιο έχει δικαίωμα προσφυγή στο ΔΕΚ και όντως με τον τρόπο αυτό υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης ε, της συνεργασίας του διαμεσολαβητή με το Κοινοβούλιο και της προσφυγής του ε, στο ΔΕΚ. Για την ε, εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Όντως είναι τεράστιο το έργο και έχω πολλά και διαφορετικά σχέδια για την εφαρμογή. Θα ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και αποδοτική αυτή η θέση. Αλλά σε περίπτωση που με εκλέξετε θα είναι πενταετής η θητεία μου θα μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Καταρχήν, να φροντίσω να υπάρχει καλή συνεργασία με τους ε, συναδέρφους μου, ώστε να τοποθετηθούν τα σωστά πρόσωπα στις σωστές θέσεις. Παρακολουθώ εδώ και 14 χρόνια τη δουλειά του διαμεσολαβητή και έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του πολύ καλά ειδικευμένου προσωπικού που έχει προσληφθεί. Δεν μπορεί να εφαρμόσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα χωρίς να υπάρχει συνέργεια και βούληση για συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Και πιστεύω εδώ ότι θα πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Θα πρέπει να προοδεύσουμε στο Βέλγιο, κανένας δεν ήθελε και κανένας δεν αναγνώρισε τον συνήγορο του πολίτη. Αναγνώριζε το ρόλο, αλλά ο διαμεσολαβητής θέλει να βοηθήσει, θέλει να βρει νέους τρόπους ώστε να αποφεληθούν όλες οι πλευρές και να εισαχθεί μια νέα φιλοσοφία στη συνεργασία. Καλή συνεργασία λοιπόν, καλό συντονισμό ανάμεσα στον διαμεσολαβητή, το προσωπικό και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι στόχος μου. Και θα ήθελα να απαντήσω αργότερα στο θέμα όσον αφορά τη συνεργασία του διαμεσολαβητή με την Επιτροπή Μεταφορών, διότι τέθηκε επανειλημμένα η ερώτηση αυτή τρεις φορές. Και θα ήθελα να ε, πω ότι είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή του ε, προγράμματός μου. Κύριε Ποστινάρο, είπαμε ότι το 75% όλων των ε, προσφυγών έχουν να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας και την άρνηση πρόσβασης στα έγγραφα. Αυτό είναι υπερβολικό. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των εθνικών συνηγόρων του πολίτη. 36% λοιπόν είναι υπερβολικό ποσοστό. Είναι ανησυχητικό, δεν θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό, αλλά είναι σίγουρα σημάδι ότι ο διαμεσολαβητής, και αυτό έχει γίνει από τους δύο τελευταίους διαμεσολαβητές τα τελευταία 14 χρόνια, ε, θα πρέπει να ε, επικεντρωθεί η δουλειά του διαμεσολαβητή στη διαφάνεια. Και βέβαια βοηθιέται ο διαμεσολαβητής από τον ε, κανονισμό 1049. Αποτελεί μία από τις δυνατότητες προσφυγών για ανθρώπου που δεν έλαβαν τι πληροφορίε που θέλουν. Μπορούν είτε να προσφύγουν στο δικαστήριο είτε στον διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, όχι μόνο για τον διαμεσολαβητή ω ε, θεσμό, αλλά και για τους πολίτες ε, να γνωρίζουν ε, ότι ε, το δικαίωμα τους στην διαφάνεια γίνεται σεβαστό. Πώς μπορεί να αυξηθεί η διαφάνεια, πώς μπορεί να μειωθεί ο αριθμός προσφυγών για έλλειψη διαφάνειας προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Συνεργασία και γνώση είναι οι απαντήσεις. Συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 1 της συνθήκης θέτει την διαφάνεια στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποθέτω ότι όπως και εγώ δεν έχετε εντυπωσιαστεί θετικά από το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον Ευρωπαίο πολίτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη διαφάνειας σίγουρα αποτελεί αιτία της έλλειψης εμπιστοσύνης. Πώς μπορούμε να ε, λύσουμε το πρόβλημα. Όλοι οι Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν καλύτερα πόσο σημαντικό είναι όχι να υπηρετούν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις, τους πολίτες. Ο πολίτης έχει αξίωση στη διαφάνεια, σύμφωνα με τη συνθήκη. Οι υπάλληλοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα. Και εγώ ήμουν υπάλληλο Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η γνώση αυτή δεν είναι αρκετά διαδεδομένη. Έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχει υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η συνεργασία. Πώς, όπως είπα στην κυρία Γκρίνη, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Μίλησα με έναν κύριο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για, όλες, για όλους τους φορείς και για τον δικό του να έχουν τη διαφάνεια στον πυρήνα των καθημερινών τους εργασιών. Δεν τον γνώριζαν αυτό αρκετό, αρκετά. Γνώση λοιπόν και συνεργασία. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, κάποιες δεσμεύσεις ε, που θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ευλογία των αρχών. Να απαντήσω στην κυρία Χάνκης. Συγγνώμη. Και εσείς με ρωτήσατε διάφορα πράγματα. Δεν θα πρέπει να ανεβάσουμε το προφίλ του διαμεσολαβητή. Δεν θέλω να επικεντρωθώ υπερβολικά στον θεσμό του διαμεσολαβητή. Επικεντρώνομαι περισσότερα στο δικαίωμα προσφυγής του πολίτη στον διαμεσολαβητή. Αυτό θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό. Με ρωτήσατε κάτι ενδιαφέρον. Μου θέσατε ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισότητα των δικαιωμάτων. Αυτό αφορά και τον διαμεσολαβητή, όχι μόνο τον διαμεσολαβητή, αλλά και αυτόν. Να, εξασφαλίσει, να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Και όσον αφορά την ισότητα, εγώ θα πήγαινα πιο πέρα. Εγώ είμαι νομικό, όπω σα έχω πει. Έχω κάνει πολλέ δημοσιεύσει όσον αφορά το θέμα τη δικαιοσύνη. Δεν είναι ακριβώ η ίδια η έννοια της ε, δικαιοσύνης στο ε, αγγλοσαξονικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο των ε, χωρών της υπηρετικής Ευρώπης, υπάρχει έννοια της αλληλεγγύης. Αυτό με έχει καθοδηγήσει στη δουλειά μου, διότι στη δημόσια διοίκηση δεν μπορούμε να ασκούμε ένα καθήκον εάν δεν διασφαλίσουμε την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Δεν έχω αρκετό χρόνο να αναπτύξω την έννοια αυτήν που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι όμως ζωτικό στοιχείο σε μια δημόσια υπηρεσία όπου ο διαμεσολαβητής έχει να παίξει έναν ρόλο, μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να γνωρίζει τα ζητήματα αυτά. Είναι αλήθεια, δεν έχω μιλήσει για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέχρι στιγμής. Και αυτό αποτελεί θέμα πυρηνικό θα έλεγα, θέμα πάρα πολύ βασικό για τον διαμεσολαβητή όπως είναι και για τον Όλαφ. Και επανέρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Γκρινή. Χαίρομαι πάρα πολύ που το νέο καθεστώς του διαμεσολαβητή του δίνει το δικαίωμα να παραπέμπει υπάλληλο στον αρμόδιο φορέα όταν καταδεικνύεται ότι ε, υπάρχει διαφθορά. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιδεινωθεί από υποθέσεις διαφθοράς. Μπορεί να έχει κανείς χίλιους υπαλλήλους απόλυτα έντιμους, μία η υπόθεση διαφθοράς να έχει κανείς. Αυτό βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πολίτες το μαθαίνουν και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώνεται λόγω αυτής της μιας υπόθεσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα διαφθοράς. αλλά η αντιμετώπιση της, διαφθορής, της διαφθοράς γίνεται εκ των υστέρων. Η κατάρτιση γίνεται εκ των προτέρων. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι να είναι απόλυτα επαγγελματικοί στον τρόπο χειρισμού των θεμάτων τους. Ελευθερία και ασφάλεια. Είναι αλήθεια ότι το ένα δεν είναι ασύμβατο με το άλλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υπάρχει μια αντίφαση. Μπορεί μπορεί στην ε, συνάντηση αυτή ελευθερίας και ασφάλειας να πρέπει να επαγρυπνεί ο διαμεσολαβητής ώστε να διασφαλίζει να υπάρχει από τη μία ασφάλεια, από την άλλη όμως να γίνεται σεβαστή η ελευθερία. Και είναι μεγάλη πρόκληση εδώ και αιώνες και θα παραμείνει η πρόκληση αυτή και τους επόμενους αιώνες. Η Ήπειρός μας έχει δημιουργήσει θεσμούς που επαγρυπνούν, που ε, καυγίζουν να το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που δημιουργούν πολιτική εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην θυσιάσουν ε, την ε, ελευθερία στο βωμό της ασφάλειας. Και αναφερθήκατε και στις παραβιάσεις εις βάρος των μειονοτήτων. Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε, να το πούμε έτσι, όσον αφορά την, την ε, ξέρω ότι ανησυχείτε για τον, ε, την προστασία των δικαιωμάτων των ε, μειονοτήτων. Στη χώρα μου το Βέλγιο υπάρχουν τρεις μειονότητες. Πολύ με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων επί εννέα χρόνια. Φροντίζω φρόντιζα να γίνονται σεβαστές οι μειονότητες. Μπορεί όμως... Μπορεί όμως να, μην είναι πάντα φιλετικές οι μειονότητες, μπορεί να είναι γλωσσικές, ε, μπορεί να έχουν να κάνουν με το φύλλο. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό θέμα για μένα επί 9 χρόνια και θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν έχω την ε, ευκαιρία, να συνεχίσω να δραστηριοποιούμε στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνεται, διότι έχουμε μείνει πίσω. Κυρία Παλιαδέλη, πώς μπορούμε να επιτυχύνουμε τη διαδικασία των ε, ερευνών. Χαίρομαι που θέσατε ερώτημα, διότι δεν θέλω απλώς να διασκορπίζω ωραίες ιδέες χωρίς να προτείνω τρόπους εφαρμογής. Αναγνωρίζω, όπως είπα εξ αρχής, ότι εγκρίθηκε το πλαίσιο ήδη και φτάνουμε στο 12ο μήνα, δηλαδή 12 μήνες είναι η μέση διάρκεια. Είμαστε στους 13, τώρα έχουμε μειώσει το χρόνο στους 12. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στους 12 μήνες που είναι και η διάρκεια που αφορά τη διαδικασία του άρθρου 226 και 228. Ο ένας χρόνος είναι αποδεκτό και σε εθνικό επίπεδο, ε, αποδεκτή διάρκεια δηλαδή. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο που έθιξα χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο ε, λύσεις με βάση τη συνένεση και απλουστευμένες διαδικασίες. Αυτό το εφήρμοσα στο Βέλγιο χρησιμοποιώντας το, τον πιο, τους πιο ευέλικτους χειρισμούς, κερδίζετε χρόνο, πολύ χρόνο, όπου εσείς και το προσωπικό σας στη συνέχεια μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στις έρευνες. Άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε πώς ε, υπάρχει, ποιο είναι το πιο ευέλικτο πλαίσιο μεταχείρισης των προσφυγών έτσι ώστε να τις εντάξουμε στις πιο παραδοσιακές έρευνες. Έτσι έχω κάνει εγώ στη χώρα μου και έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Χάρκιν, κυρία Χάρκιν, όχι Όκεν, Χάρκιν, συγγνώμη γιατί κακοπρόφερα το όνομα. Μου υποβάλλετε μια σειρά ερωτήσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο κατανόησα αυτό το πρώτο ερώτημα σε σχέση με τις ε, νέες προκλήσεις και τα παραδοσιακά δικαιώματα. Ως προς το δεύτερο ερώτημα σας, η Ευρώπη βασίζεται στο common law, στο αγγλοσαξονικό σύστημα από την ε, άλλη πλευρά, το common law και το equity law, που είναι το αγγλοσαξονικό και το υπηρετικό δικαιοδοτικό σύστημα από την άλλη. Νομίζω ότι πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιοδοτικά συστήματα. Όπως είπα και στην κυρία Χάνκης, στο Βέλγιο χρησιμοποίησα το equity law για να το εισαγάγω στο δικό μας νομικό σύστημα, στη δική μας χώρα. Και ήταν πολύ δύσκολο να πείσω το Κοινοβούλιο, τους ε, ορίζοντες τις πολιτικές και τους ακαδημαϊκούς ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι μια αρχή που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το νομικό μας σύστημα. Γι' αυτό πιστεύω στο συμπληρωματικό χαρακτήρα των δύο συστημάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο και στα δύο συστήματα στον τρόπο χειρισμού των ε, προσφύγων. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναπτύξω, αλλά δεν έχω χρόνο, είναι ότι στην Ευρώπη γνωρίσαμε τρεις ε, γενναίες ομπούτσμεν. Ε, δεκαετία του 70, η πρώτη γενναία στις σκανδιναβικές χώρες, μετά τις δικτατορίες σε πολλές χώρες και μετά την κατάρριψη του τείχους. Αυτές οι γενές ombudsman δημιούργησαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Όλα τα συστήματα είναι χρήσιμα γιατί είναι συμπληρωματικά. Και αυτό είπα και εγώ. Γιατί θα πρέπει κανείς να είναι ombudsman για ολόκληρη την Ευρώπη μέσα στα πλαίσια των δύο συμπληρωματικών συστημάτων, συμπληρωματικών κατά τη γνώμη μου. Πώς ορίζω την κακοδίκηση όταν ο κύριος Σέντερμαν, ο πρώτος ομπουτσμαν, πρότεινε στο Κοινοβούλιο Έχω την επιστολή που του είχα γράψει τότε, νομίζω το 96-97, όταν ε, του ζητήθηκε ο ορισμός της κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης, είπε ότι θα πρέπει να καλύπτει την παραβίωση ενός δεσμευτικού νόμου ή αρχής και ήδη 14 χρόνια πριν διαφώνησε και το έγραψα όχι. Θα πρέπει να είναι ευρύτερος ο ορισμός. Η κακοδίκηση πρέπει να περιλαμβάνει τις παραβιάσεις του ήπιου νόμου μια αρχής, ακόμα και αν δεν είναι δεσμευτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κακοδιοίκηση σημαίνει παρανομία. Κακοδιοίκηση δεν σημαίνει υποχρεωτικά παρανομία. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε μια ευρύτερη ενιολογική βάση ως προς τον ορισμό. Τώρα θα ήθελα να, ερωτήσω, να απαντήσω σε ερωτήσεις που μου θέσατε ως προς συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Πιστεύω, επειδή παρακολούθησα την ιστορία αυτού του θεσμού, νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Ombudsman, είδαμε τον κύριο Σέντερμαν, τον κύριο Διαμαντούρο, Στη συνέχεια η συνεργασία ήταν αγαστή με την Επιτροπή Αναφορών. Έχει βελτιωθεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν επικρίνω τίποτα οι άλλες χώρες. Πιστεύω όμως ότι η συνεργασία είναι πολύ καλύτερη από ότι σε συνεργασία εθνικού επίπεδου. Ίσως ε, είναι ένα παράδειγμα προς από εθνικούς ε, συνηγόρους του πολίτη. Αυτό που είπα και η κυρία Παλιαδέλη είπε ακριβώς το ίδιο, είναι ότι για, σε θέματα επικάλυψης μεταξύ Ombudsman και Επιτροπής Αναφορών θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο για να μην έχουμε την, το διπλό φόρτο. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε ολοένα και περισσότερο να βρούμε ζητήματα ή προσφυγές όπου οι αναφορές αφορούν ε, μία συλλογική προσφυγή όπου ο Ομπούτσμεν ήταν δραστήριος και ίσως θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών και επικοινωνία γενικά όταν εργαζόμαστε σε παρόμοια ζητήματα. Τώρα, κυρία Άουκεν, κυρία Όκεν, μου υποβάλατε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα νομικής υφής. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί ή δικαιούται, ας το πούμε έτσι, να αποτιμήσει τον τρόπο που έχει χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τα άρθρα 226 και 228, η χρήση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπα ότι σε διαδικαστικά αλλά και σε θέματα ουσίας μπορούμε να κρίνουμε την χρήση, την κατάχρηση, την έλλειψη χρήσης αυτών των αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Δεν λέω ότι ο ομπουτσμαν θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτές τις δικαιοδοσίες του 226-228 το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαίου Ομπουτσμαν και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δύο αυτά άρθρα ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διακριτική ευχέρεια χρήσης ημί του 226 και η διακριτική αυτή ευκαιρία μπορεί να επικριθεί, αλλά έχει ε, εγκριθεί από το ΔΕΚ, άρα δεν τίθεται εν κινδύνο. Άρα λέω ότι ο Ομπούτσμαν ήδη λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αν διαβάσετε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, βλέπετε ότι έτσι κινείται σε διαδικαστικά ζητήματα ή σε θέματα ουσίας για την εφαρμογή του 226. Ο Ombudsman μπορεί να ορίσει ότι η Επιτροπή δεν έκανε λογική χρήση του 226. Και τώρα στρέφουμε σε μια βασική αρχή που έχει αναπτυχθεί στο Βέλγιο, το θέμα του ευλόγου. Δηλαδή, κατά πόσο ένας φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εξουσία και δεν μπορεί να την ε, ε, χρησιμοποιήσει εφόλου της ύλης. Δηλαδή, η διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά. Και αυτό αφορά διάφορα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα. Δηλαδή, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της, αλλά με βάση μια ορθολογική χρήση όπως ισχύει και στην περίπτωση του διαμεσολαβητή, ο οποίος ξέρει ή θα πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο το 226 ή 228 έχουν χρησιμοποιηθεί εύλογα. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί ορθολογικά αυτά τα δύο άρθρα ή έχουν ε, ή, ε, ή, έχει γίνει κακή χρήση. Ο κύριος Σαλαβράκος έχει φύγει, αλλά θα το απαντήσω. Είπα ότι δεν υπάρχει καμία ένταση μεταξύ της ε, δικής σας Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εδώ και 14 χρόνια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μια στενότερη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αρχίζει η διαδικασία του Catch the Eye. Εντάχει μόνο ένα αίτημα έχω από την κυρία Χάπινγκ και θα της δώσω ένα λεπτό καθώς και ένα λεπτό για την απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω Ολλανδικά γιατί και ο μιλητή μα μιλάει τόσο καλά ολλανδικά. Ακούγοντα λοιπόν το πρόγραμμά του μου φαίνεται τόσο φιλόδοξο όσο και του Ομπάμα. Πώς θα γίνει όμω αυτό, γιατί βρίσκεται σε μία απομόνωση στο Στρασβούργο. Εγώ εργάστηκα στο γραφείο του Επιτρόπου Κάλλας και ήμουν ο αντίθετος πόλο αν θέλετε, του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στο γραφείο αυτό και συχνά αναζητήσαμε φιλικές λύσεις. Συμφωνούσαμε τον ε, διαμεσολαβητή, αλλά η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπαν ότι «Α, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται για τον τάδε ή δίνα λόγο» και υπήρχε μια έντονη, αν θέλετε, ε, προάσπιση της, των δικαιωμάτων του διαμεσολαβητή. Ήταν αρκετά άκαμπτη η στάση του. Σας ρωτώ λοιπόν πώς θεωρείτε ότι θα διαμορφωθεί ο ρόλος σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί είπατε ότι θέλετε να δραματίσετε ιδιαίτερα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα διαφημίσετε στον τύπο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι αν εκλεγείτε κάθε επιτυχία σε ό,τι αφορά την μεταρρυθμιστική σας αυτή ατζέντα που θυμίζει ο Ομπάμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου ταιριάζει πολύ με αυτά που είπε ο προλαλή σα. Όταν ακουστεί, όταν οι πολίτες της Ευρώπης έχουν την εντύπωση, λάβουν την εντύπωση ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να κινήσει πολλά, τότε και οι προσφυγές θα αυξηθούν. Αν υπάρχει εντύπωση ότι δεν έχει κανένα νόημα, τότε δεν προσέγγει κανείς το διαμεσολαβητή. Πολύ ωραία ακούγεται και το υπογράμμισα ότι το πιο σημαντικό είναι να μην διαρκεί πολύ η προσφυγή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι Τι θα πρέπει νομοθετικά να αλλάξει για να αυξηθεί η βελτίωση και χρειάζεστε τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να πολεμήσουμε σε όλα τα μέτωπα και εμείς έχουμε το στόχο τις αναφορές να τις επεξεργαζόμαστε γρήγορα. Διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα σε μια απάντηση και μάλιστα δικαίωμα σε απάντηση μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι το, το ερώτημά μου. Κύριε Επίνκ, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή που μου θέσατε. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξο το πρόγραμμά μου. Δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κανείς φιλόδοξος σε μια τέτοια θέση. Όντω είπα ότι ασχολούμαι εδώ και χρόνια στο πλαίσιο διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρω πόσο δυνατά μπορεί να είναι τα θεσμικά αυτά όργανα για την υπονόμευση μεταρρυθμίσεων. Όντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα, παρουσιάζονται κατά καιρούς ε, παραδείγματα θεσμικά όργανα, υπάλληλοι οι οποίοι δεν είναι υπέρ των αλλαγών. Αυτό όντως αληθεύει. Αλλά αυτό αποτελεί και τμήμα, αν θέλετε, της καθημερινότητας των θεσμικών οργάνων και σε εθνικό επίπεδο είναι καθημερινό φαινόμενο ότι ο μεσολαβητής, ο συνήγορος του πολίτη, να ζητά διαρκώς αλλαγές, να ζητά διαρκώς πιο πολύ διαφάνεια, πιο πολύ ανοιχτό χαρακτήρα και επί εννέα χρόνια ασχολούμαι με τέτοια ζητήματα. Ασφαλώς και τα πράγματα δεν γίνονται σε μία νύχτα. Και έμαθα να είμαι υπομονετικός αλλά και επίμονος. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να επιτυχάνονται οι στόχοι μας. Αυτά δεν συμβαίνουν σε μία νύχτα, όπως είπα. Μου θέσατε και μια δεύτερη ερώτηση για το πώς θα προβάλλω το έργο μου, το έργο των συνεργατών μου στον τύπο, στο ΜΜΕ. Να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα διάφορα χώρα, διάφορες χώρες. Τη Γαλλία, το Βέλγιο και το καθεξής. Όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συμφωνίες με τον τύπο για να γνωρίσουν καλύτερα τα μέσα τη λειτουργία των θεσμικών αυτών ε, θέσεων. Δεν, είναι, δεν μιλάω απαραίτητα για συνέντευξη τύπους, τύπου, αλλά γενικά δράσεις για την προώθηση της ε, ευκρίνειας, αν θέλετε, του έργου του κάθε θεσμού. Δεν έχω πολύ χρόνο να απαντήσω στον επόμενο ομιλητή, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να γεννηθεί μια ελπίδα στον κάθε πολίτη αν δεν γίνεται σεβαστή η ελπίδα αυτή. Συμφωνώ απόλυτα και... Το έχω ζήσει, το έχουμε δει στο Βέλγιο, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Όντως αληθεύει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και είπα ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε. για να γίνει πιο γνωστό το δικαίωμα του πολίτη να αποτανθεί στον διαμεσολαβητή και να αναπτυχθούν σχετικά προγράμματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν προσφεύγουν στο διαμεσολαβητή για θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα χωρίς το άλλο. Θα ήταν πραγματικά τρομακτικό. Θα πρέπει να υπάρχει η σωστή συνεργασία στο επίπεδο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μονέτ. Έληξε η ακρόαση. Σας χαιρετούμε. Έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε με τις εργασίες μας. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή δεν έχει ούτε καθήκον ούτε εξουσία να αποφασίσει ή να ε, εκφράσει απόψεις μετά από αυτό το μαραθώνιο. Μπορούμε απλώς να διαβάσουμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τα πρακτικά αυτών των ακροάσεων με όλες τις παρεμβάσεις και τις επεξηγήσεις ως προς τις τρεις αυτές ακροάσεις ε, των τριών υποψηφίων. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις ή υποδείξεις, θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίαση με τη δέσμευση να διαβιβάσουμε στον